All right. Colleagues, may I have your attention, please? Πρόεδρος, συνάδελφοι, παρακαλώ, προσέξτε και καθίστε. Έναρξη της συνεδριάσεως. Και πρώτα πρώτα, να σας ζητήσω συγγνώμη. On her way to this meeting, and uh, we felt that we should not. Κύριε Μπόλς, κάπου με το χιόνι κάπου κόλλησε. Οπότε και εγώ προσφέρθηκα να προεδρεύσω μέσω του η πρόεδρος μας ή κάποιος αντιπρόεδρος άλλος έρθει να προεδρεύσει. Πρώτα πρώτα ε, κάνουμε την έγκριση της μεσαίας διατάξεως. Αν δεν έχετε κάποια ένσταση, ε, κάποια τέλος πάντων πρόταση, τότε θεωρώ ότι εγκρίνεται. Επίσης, σας ενημερώνω ότι έχουμε εδώ μια σειρά πρακτικών από την αρχή Νοεμβρίου μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, τα οποία έχουν αποκρισταλωθεί και αν δεν έχετε αντίρρηση θεωρώ ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Επίσης έχω μια σειρά ανακοινώσεων που καλύτερα η κυρία Μπούλ να σας τα πει. κάποια στιγμή. Αργότερα σήμερα, αύριο το πρωί, αύριο το απόγευμα, κάποια στιγμή. Και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό. Για σήμερα το απόγευμα είναι τιμή μα να υποδεχόμεθα εδώ τον κύριο Βιτόριο Γκρίλη, Υπουργό Εθνική Οικονομία Οικονομών τη Ιταλία. Μπενβενούντο. Και σα ευχαριστούμε που ήρθατε. Διαφέρομαστε πάρα πολύ να μας πείτε πώς αποτιμάτε την κατάσταση η χώρα σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Παρακαλώ, όπως έχουμε πει, θα κάνουμε μια ε, εισήγηση δεκάλεπτη και κατόπιν ε, θα υπάρξει το περιθώριο για τους συναδέλφους, τους ευρωβουλευτές, να σας ε, υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Ακριβώς όπως έχουμε ήδη συμφωνήσει. Και Βέβαια, δεν είναι δικό μου θέμα να κάνω την ε, σύνοψη σε σχέση με το τι κατάσταση επικρατεί σήμερα στη χώρα σας. Αυτό το κάνετε εσείς, είστε εσείς, να το κάνετε πολύ καλύτερα από μένα. Και κατόπιν, αυτής αμέσως τώρα θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκρίλη. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Οικονομικών Υποθέσεων, μεγάλη μου χαρά που σήμερα παρίσταμε εδώ, εμφανίζομαι ενώπιόν σας εδώ, στα πλαίσια του οικονομικού διολόγου. Δέκα λεπτά είναι πάρα πάρα πολύ λίγα. Για να μπορέσω να σας παρουσιάσω το θέμα μου. Και βέβαια, όταν έρθει η ώρα των ερωτήσεων, θα έχω την ευκαιρία να σας πω λεπτομέρειες να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη πιο συγκεκριμένα. Θέλω να σας τα πω στα Ιταλικά, την δική μου γλώσσα, για να σας πω το πώς έχει κατάσταση στη δική μου χώρα. Μετά από μία σειρά μηνών εντάσεων, τώρα στην Ευρωζώνη τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, βελτίωση όλων των μεταβλητών, τα spreads, οι ροές των κεφαλαίων, καταθέσεις παντού, σε όλες τις τράπεζες και όλα δείχνουν ότι η κατάσταση βελτιώνεται στις αγορές. Χρηματοοικονομικές συνθήκες, επομένως που έχουν τώρα βελτιωθεί, διασκεδάζουν τους φόβους για τις προοπτικές της Ακόμα όμως η κρίση δεν τελείωσε. Όμως Νομίζω ότι η συγκυρία είναι καλύτερη και επομένω νομίζω ότι πρόκειται για μια κρίσιμη, καλή, ευχάριστη καμπή, ώστε τα πράγματα πάνε καλύτερα το δεύτερο ημίση του 2013. Οπότε, βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τόσο ικανοποιημένοι. Ο ρυθμός της ανάπτυξης είναι τέτοιο που δεν μπορούμε ακόμα να φτάσουμε στη κατάλληλη απασχόληση που θέλουμε και έτσι επομένως έχουμε τέτοιες προοπτικές Οπότε θα πρέπει τώρα να λάβουν όλα τα κράτη-μέλη τι ευθύνε του και επίση όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Χρειάζεται μια αναδιάρθρωση βαθιά. Έχει ξεκινήσει ήδη σε μια σειρά χωρών, οπότε να εφαρμοστούν όλα τα σχετικά με την δέουσα μεταρρύθμιση. Τα πράγματα είναι κοινωνικά δύσκολα, πολιτικά δύσκολα, αλλά έτσι θα πρέπει να δούμε πώς θα φτάσουμε στα υποθητά αποτελέσματα. Ότι μέλη και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεχίσουν την κοινή γραμμή για την ε, διακυβέρνηση και κατά τη γνώμη μου. Έτσι, έχουμε βελτίωση το των με αυτό, αντικατοπτρίζει το τι γίνεται με τα θεσμικά όργανα, με τα κράτη-μέλη, τα οποία μπόρεσαν να έχουν κάποιο είδου αξιόπιστη και αποτελεσματική στρατηγική ενάντια στην κρίση. Τα, τα πρόσφατα χρόνια, το 2012, είχαμε σημαντικές αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν και είχαμε θαραλέε επίση ε, κινήσει κατόπιν των όσων αποφάσισε τελείω Ιουνίου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο. Επομένως αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να σταματήσει ε, αυτός ο φαύλος κύκλος ε, με το, το, τα χρέη και το έλλειμμα, οπότε έχουμε αυτόν τον ε, μηχανισμό σταθερότητας και έτσι να μπορέσουμε, είπαμε, να μπορέσουν οι χώρες και οι γλώσσες να έχουν προσβασιμότητα σε αυτό το ταμείο και είπαμε επίσης ότι και η κεντρική ε, τράπεζα μπόρεσε να βοηθήσει όσον αφορά τον φόρο των συναλλαγών και έτσι εδώ συγκρατήσαμε τον κίνδυνο παντού στην Ευρώπη. Και γι' αυτό λοιπόν και αμυφθήκαμε με την αύξηση τη αξιοπιστία μα. Επίση, πρέπει να έχουμε έναν ενιαίο επιτοπτικό μηχανισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτω ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την ιδέα τη Τραπεζική Ένωση, όπω δεν προανέφερα. Η πρόοδο αυτή σημειώθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά επίσης και σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, επιτρέψτε να σας υποβάλω κάποιες παρατηρήσεις για τη δική μου χώρα. Αλλά τώρα θα σας τα πω στην εθνική μου μητρική γλώσσα. Στην Ιταλία τα σε εθνικό επίπεδο μάλλον τα κράτη-μέλη έκαναν μια προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης με συνοδεία μεταρρυθμιστικών πολιτικών για να αντισταθμίσουν την αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη. Η Ιταλία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ε, έγινε μια θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πέρυσι. Η Ιταλία έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες ε, μεταρρυθμίσεων και σταθεροποίησης. Η κατάσταση στο προϋπολογισμό μας είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι σε άλλες ε, αναπτυγμένες χώρες. Παρ' αυτά υπήρξε κρίση εμπιστοσύνη στις αγορές και αυτό ε, έπληξε την Ιταλία. Έτσι έχουμε μπει σε μια φάση ύφεση πιο μεγάλη από ό,τι περιμέναμε. 2,4% ε, μειώθηκε η ανάπτυξή μας, αλλά το πρώτο εξάμεινο του 2013 θα σταματήσει αυτή η ύφεση και θα έχουμε ανάπτυξη επόμενη, το επόμενο, ε, την επόμενη μισό του 2013 τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μία ανάπτυξη 1% ε, από το 2014 και τα λοιπά. Η ανάπτυξη λοιπόν της οικονομίας μας θα προωθηθεί χάρη σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων. Εδώ σημαίνει το μεταρρύθμιση στο σταξιωτικό σύστημα, στην αγορά εργασίας, ε, αποτελεσματικότητα στο δημόσιο τομέα. Αυτά τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει, ε, θα έχουν σκοπό να επιτύχουμε μία ανάπτυξη 4% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, τα μέτρα που υιοθετήσαμε ε, έχουν σκοπό να οδηγήσουν σε ανάπτυξη του ΑΕΠ περίπου 3%. Ε, σε σχέση με το 12 ε, και μέχρι το 15 θα φτάσει στο 5%. Εμείς έχουμε φέτος μείωση του ΑΕΠ κατά 1%. Αλλά ήδη θα έχουμε μία ανάπτυξη από το δεύτερο μισό του 2013, όπως σας είπα. Η κυβέρνηση έχει μετακινήσει τη φορολογία από την, από την εργασία και τον κατασκευαστικό τομέα έχουμε ένα πακέτο μέτρων για να προωθήσουμε την, την καινοτομία, να ευνοήσουμε την ανάπτυξη και να μειώσουμε σε ορισμένου τομεί την φορολογία για να προωθήσουμε την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και να τις, τους δώσουμε τα καλύτερα μέσα για να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η, η Ιταλία αλλάζει, αλλάζει βαθιά το 2012 το κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο μας ε, ενέκρινε μια τροπολογία ε, για να εισαγάγει την έννοια του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού που θα είναι μια προϋπόθεση θεσμευτική από το 2014 και αφορά ολόκληρο το δημόσιο τομέα. Αυτή η αρχή λαμβάνει υπόψη τις κυκλικές αλλαγές και τις έκτακτες συνθήκες μέσα στις οποίες ε, τις οποίες ζούμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ιταλικό Κοινοβούλιο ε, υιοθέτησε και ένα νομοσχέδιο, το λεγόμενο ενισχυμένο νόμο, ούτω ώστε να έχουμε εξισορρόπηση του προϋπολογισμού και θα υπάρχει και ένα μας ανεξάρτητος φορέας ο οποίος θα ε, ελέγχει το φορολογικό και τη δημοσιονομική κατάσταση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα για την σταθεροποίηση του προϋπολογισμού, αλλά κάναμε και πολλές άλλες πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές δράσεις. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω μόνο κάποια από αυτά τα μέτρα και μετά θα σας δώσω το λόγο, ούτως ώστε να μπούμε σε μια πραγματική συζήτηση. Κάνουμε παρεμβάσεις για τη διαφάνεια και την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχουμε μια επιτροπή για την αξιολόγηση ακριβώς ε, της, της ε, διαφάνεια στο δημόσιο τομέα. Θα είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, μεγαλύτερη διαφάνεια και της ε, γραφειοκρατίας μας. Προβλέπουμε την δημοσίευση σε ιστοσελίδες όλων των εργασιών της δημόσιας διοίκησης, όλων των διοικητικών αποφάσεων που αφορούν και τον προϋπολογισμό, αλλά και οποιαδήποτε δημόσια έργα. Επίσης, ε, η καταπολέμηση της διαφθοράς ε, διευκολύνεται και ενισχύεται μέσω πιο αυστηρών ποινών για τους δημόσιους λειτουργούς. Επίσης, το ελεκτικό μας συνέδριο έχει περισσότερες εξουσίες για να ελέγχει τους προϋπολογισμούς των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των δήμων, κοινοτήτων κτλ. Επίσης, διαδικασίες απλουστευμένες για έργα υποδομής. Ε, αυτό ξεκίνησε να ισχύει το τελευταίο τρίμηνο. Ξαναείδαμε τους ε, δημοσιονομικούς ε, και χρηματοοικονομικούς κανόνες και για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Επίσης, από την αρχή του 2013 οι πληρωμές ανάμεσα στον, στο δημόσιο τομέα προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 30 μέρες. Επίσης, μετά από τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας πέρυσι, οι εργοδοτικές οργανώσεις έφτασαν σε μια συμφωνία με την κυβέρνηση, ούτω ώστε να προωθήσουμε συμβάσεις ε, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και για να ενθαρρύνουμε αυτή την αλλαγή, η κυβέρνηση έχει προωθήσει πόρους 2,1 ε, εκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, που θα πάνε σε μέτρα ε, για την αντιστάθμιση πιθανών θέσεων απασχόλησης. για την αντιστάθμιση της απώλειας πιθανών θέσεων απασχόλησης. Εν κατακλείδη θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει μία διαδικασία, μία πορεία. Η κυβέρνηση έκανε μια αποφασιστική προσπάθεια. Φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ η προσπάθεια όλα τα υπεύθυνα θεσμικά όργανα και οι φορείς σε εθνικό επίπεδο θα συνεχίσουν αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που ξεκίνησε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, για τη σύντομη αυτή παρουσίασή σας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση. Ξέρουμε όλοι ότι η Ιταλία κυβερνάται σήμερα από μια κυβέρνηση γραφειοκρατών, εμπειρογνωμόνων. Ξέρουμε ότι η χώρα σας την άλλη τον άλλο μήνα θα έχει εκλογές και φαντάζομαι ότι κάποια από τα ερωτήματα που θα σας απευθυνθούν θα έχουν να κάνουν και με το πολιτικό μέλλον της χώρας σας. Τώρα, συνάδελφοι, ξέρετε όλοι τι μορφή θα ακολουθήσει η συζήτηση. Έχουμε πέντε λεπτά ο καθένας για ερώτηση και για απάντηση. Άρα, όσο πιο πολύ, όσο λιγότερο χρόνο Πάρατε με την ερώτηση, τόσο πιο πολύ χρόνο θα έχει ο Υπουργό για να απαντήσει. Αν μπορείτε λοιπόν, περιοριστείτε σε ένα 1,5 λεπτό. Ο Ζαν Κοζέ εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Υπουργέ, στη συνεδρίαση τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Θα σα θέσω μια αφελή ερώτηση που τη θέτουν και οι πολίτε. κάτι που σχετίζεται με αυτά που είπατε στην αρχή για την Ευρωζώνη. Πώς γίνεται μέσα τόσο λίγο χρόνο, τη στιγμή που κανένα από τα μέτρα που δεν έχουν προναγγελθεί έχει εφαρμοστεί ακόμα, όλα είναι σε φάση συζήτηση. πώς γίνεται έφνης κάτι γνώμη σα, οι αγορές να αλλάζουν και ενώ επί χρόνια λέγανε ότι είμαστε στο χείλος καταστροφής εμείς η Ευρωζώνη, ε, συζητήσεις, ε, φασαρία κτλ. Πώς γίνεται μέσα σε λίγου μήνε ενώ τίποτα πραγματικά δεν έχει υλοποιηθεί, πώς εξηγείται ότι η εκτίμηση για την Ευρωζώνη έχει αντιστραφεί εντελώ. Μπορείτε να μιλήσετε και για την Ιταλία, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάντω. Ευχαριστώ. Δεν συμφωνώ 100% με την υπόθεσή σας, ότι τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Θεωρώ ότι οι αγορές κοίταζαν και κοιτάζουν με πολύ προσοχή την εξέλιξη και σε επίπεδο διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, αλλά και την κατάσταση στις επιμέρους χώρες. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι αποφασιστικά. Και ακριβώς δείχνω ότι υπήρξαν εφαρμογές των μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε μια σημαντική συμφωνία για το ESM, όπως και η προαναγγελία της Κεντρικής Τράπεζας, των μέτρων που θα πάρει, όλα αυτά τα μέτρα δεν χρειάζεται να εφαρμοστούν κατά ανάγκη. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν. Ε, είναι μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το σύστημα εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Αυτά τα πήραμε σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα όλα αυτά τα μέτρα. Και οι αγορές κατάλαβαν την αποφασιστικότητά μας, των κρατών μελών δηλαδή και των θεσμικών οργάνων, για να κάνουμε κάτι. Επίσης κατάλαβαν ότι μπορούμε να αποφασίσουμε και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους ε, χώρες, μόνο για την Ιταλία εγώ μπορώ να μιλήσω προφανώς. Φέτος, πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που πέρασαν από το Κοινοβούλιο εισήχθησαν και εφαρμόζονται. Ένα παράδειγμα η πολύ σημαντική φάση ολοκλήρωσης ε, του της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως σας είπα έφτασε σε τελεσφόρηση, ξεκίνησε με μια νομοθετική προσπάθεια. Και εφαρμόζεται αυτή η μεταρρύθμιση χωρίς να χρειαστούν περαιτέρω διοικητικές αποφάσεις ή μεταρρυθμίσεις, κάτι που είναι πολύ θετικό. Όταν ξέσπασε η κρίση, σε μεγάλο βαθμό ήταν μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην Ευρώπη και στην ικανότητά της να εξελιχθεί και να ανταποκριθεί στην κρίση. Ήταν μια κρίση που αφορούσε και τις προσδοκίες. Προσδοκίες που είχαν οι αγορές από τις επιμέρους χώρες και από την Ευρώπη, αλλά και την Ευρωζώνη πιο συγκεκριμένα, να ότι μπορούν να αντιδράσουν ε, με συγκεκριμένα εργαλεία και μέσα για να ανταποκριθούν, για να απαντήσουν σε αυτή την κρίση. Ξέραμε, μάθαμε και είδαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε. Και αυτές οι προσδοκίες που ήταν προβληματικές στην αρχή έγιναν θετικές και τώρα βλέπουμε ότι οι αγορές ξαναβρίσκουν την εμπιστοσύνη τους στην Ευρώπη, στα κράτη-μέλη, ότι μπορούν να αντιδράσουν και ότι μπορούν να δώσουν αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα χρονοδιαγράμματα με ορόσημα, συγκεκριμένες προθεσμίες και μέσα στην τελευταία χρονιά, 1,5 χρόνο, είχαμε πολλές προσπάθειες επίλυσης της κρίσης στις διάφορες χώρες, μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Είχαμε αναγγελίες συγκεκριμένων προγραμμάτων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και αυτό είχε θετική απήχηση. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ο κύριο Πιτέλα, για τους e grazie. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την ανοιχτή σας τάση και την ε, ζεστή αντιμετώπιση του Κοινοβουλίου. Την περασμένη Παρασκευή η Τράπεζα της Ιταλίας για το 2013 ανήγγειλε μία μείωση της ανάπτυξης. Έχουμε σύμπηξη του ΑΕΠ του 0,2 ΑΕΠ. Είναι πολύ δύσκολο, λοιπόν, μέσα με αυτές τις κακές προβλέψεις να εξισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. Έχω δύο ερωτήσεις. έχουμε απτά αποτελέσματα της λιτότητας. Δεν θα πρέπει επομένως να βάλετε κάποια όρια ε, στα μέτρα λιτότητας για να μην επιδεινωθεί η κοινωνική κατάσταση της χώρας. Επίσης θα ήταν πιο σωστό να πείτε ότι λόγω του ότι έχετε, έχουμε τόσο προβληματική κατάσταση στην Ιταλία, ε, είναι αδύνατον να φτάσουμε σε εξισορρόπηση του προπολογισμού μέσα στο 2013. Ε, κάτι που αποφασίστηκε, που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση Μπερλουσκόνη με τρόπο α, ανεύθυνο θα έλεγα. Έχω να απαντήσω καταρχήν καταφατικά στην ερώτησή σας. Αλλά κοιτάξτε τι έκανε αυτή η κυβέρνηση. Ε, η εξοσκέληση του προϋπολογισμού του 2013 ε, δεν είναι ονομαστική εξισορρόπηση, αλλά αφορά τις δομές. Δηλαδή, όταν το Δεκέμβριο του 2011 κάναμε αυτή την ε, διορθωτική προσπάθεια για να εξοσκελίσουμε τον προπολογισμό, οι τότε οικονομικές προβλέψεις ήταν πιο ευνοϊκές, ήταν διαφορετικές από αυτές που έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν ε, οι προβλέψεις ε, της Τράπεζας της Ιταλίας ε, συμπίπτουν με τις ε, κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή κατάσταση είναι τελείως διαφορετική από την κατάσταση του 2011, είναι χειρότερη. Αυτό το ξέραμε και την περασμένη Άνοιξη. Εμείς ως Ιταλία, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθορίσαμε μια αρχή πολύ σημαντική. Δηλαδή, ότι δεν θα προσφύγουμε, δεν θα επιμείνουμε στην ύφεση. Δηλαδή, όταν εμείς κάναμε το Δεκέμβριο του 2011 ε, αυτό το διορθωτικό νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, ε, είχαμε σαν σκοπό ε, την διαρθρωτική αλλαγή, όχι την ονομαστική αλλαγή. Δηλαδή, για το 2013 δεν είπαμε θα πρέπει να έχουμε απόλυτη ισορροπία, αλλά θα πρέπει να έχουμε εξισορρόπηση μετά από όλες τις προσαρμογές και τις κυκλικές αλλαγές. Εάν αυτό το 0,2% επιδεινωθεί, αυτό θα απεικονιστεί και στο στόχο μας για τον προϋπολογισμό. Αυτά που λένε οι εφημερίδες δεν είναι σωστά. Ο στόχος είναι να, προσαρμόσουμε, να προσαρμοστούμε στην ε, φάση του οικονομικού μας κύκλου, δηλαδή να τη λάβουμε υπόψη μας κατά την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε επιπλέον την οικονομία σε μια τόσο δύσκολη στιγμή με επιπλέον μέτρα λιτότητας. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ε, της ε, ισοσκέλησης του προϋπολογισμού. Και ακόμα τα ίδια λέμε και, στην, ε, και στο Δούνου του. Θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή κυκλική αναπροσαρμογή. Και αυτήν τη συμπεριλαμβάνουμε στα νούμερα τα οποία δημοσιεύουμε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Είμαι καταλανός ε, ευρωβουλευτής και θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Χθε το βράδυ ο, ο κύριος Μόντι μίλησε για τις βαθιές μεταρρυθμίσεις στην Ιταλία. Ποιε είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα λάβουν χώρα πέρα το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια που δεν έχουν γίνει ακόμα. Υπάρχει περίπτωση επίσης να γίνει α, μεταρρύθμιση στις περιφέρειες όπως έγινε ας πούμε στη Γερμανία, ούτως ώστε να μην ξοδεύουν οι περιφέρειες χρήματα, αλλά να υπάρξει μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Θα πρέπει να απαντήσω σε δύο επίπεδα. Πρώτον, αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε τα διαρθωτικά προβλήματα της Ιταλίας, δηλαδή τα ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, με πλήρη και ευρύ τρόπο. Υπήρχαν όμως τομείς που η κυβέρνηση δεν άγγιξε καθόλου. Είναι σωστό και λογικό να πούμε ότι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν πάνε σε βαθύ επίπεδο. Χρειάζεται μια προοδευτική και συνεχή δράση η Ιταλία. Σε ορισμένου τομεί των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη εισαχθεί, πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερο βάθος. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διάτρηση σε ένα χιλιόμετρο ε, σε βάθος, ε, σε ορισμένες περιοχές, ενώ σε άλλους τομείς θα πρέπει να πάμε πιο επιφανειακά. Δηλαδή δεν πρέπει να αγγίξουμε πιο πλατιού πιο πλατιούς τομείς, αλλά να πάμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ε, μερικά πράγματα πρέπει να τα βάλουμε βαθμιδών και όχι με μια. Υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μεταγενέστερα βήματα, κυρίως στο δημοσιονομικό πλαίσιο, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την σταθερότητα των δημόσιων λογαριασμών. Ειδικά, σε, ειδικά μεσοπρόθεσμα, Έχουμε ήδη πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την δημοσιονομική σταθερότητα. Ε, έχουμε προβλέψει το κόστος των συντάξεων κτλ. Υπάρχουν άλλα, άλλοι τομείς όπου πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω σε μεγαλύτερη εμβάθυνση, μεγαλύτερη απελευθέρωση ε, και εξασφάλιση μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας της ιταλικής οικονομίας. Κάτι που περνάει μέσα από την αναπροσαρμογή του δημόσιου τομέα. Ο δημόσιος τομέας. Πρέπει να δούμε καταρχάς τη διάστασή του, τις διαστάσεις του και το σχεδιασμό του. Τις σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στις ε, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Ο σχεδιασμός που κληρονομήσαμε ίσως δεν είναι ο ιδανικός. Η δική μου κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό έστειλε μια πρόταση συνταγματικής μεταρρύθμισης στο Κοινοβούλιο πριν από λίγους μήνες, ούτω ώστε για να δούμε, να δούμε ποιες είναι οι εξουσίες, ποιες είναι οι αρμοδιότητες των περιφερειών και του κράτους. Κάνουμε καλύτερο, μια καλύτερη διαίρεση των αρμοδιοτήτως ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των περιφερειών στο εξωτερικό, ε, τον τρόπο που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Σε ό,τι αφορά την ε, δημοσιονομική ευθύνη, που συνδέεται με την ε, ευθύνη για τις δαπάνες. Έχουμε κάνει πράγματα Έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόσουμε ένα μέτρο το 2011. Να ξαναδούμε τη φορολογία για τα κίνητα. Αλλάξαμε τη φορολογία στα ακίνητα. Ήταν σχεδιασμένη η φορολογία αυτή ως ένα σύνθετος φόρος. Εν μέρη πήγαινε στο κράτος και εν μέρη πήγαινε στις τοπικές αρχές. Τώρα αλλάξαμε το σχεδιασμό αυτού του φόρου. Πηγαίνει ε, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων στις ε, τοπικές αρχές και είναι και ένα από τα μεγαλύτερα εσόδά τους. Έτσι λοιπόν έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια, αλλά θα πρέπει αυτή να, να την παγιώσουμε και μέσα από μια ε, μεταρρύθμιση του συντάγματος. Φίλιπ Λάμπερτς the... από τους Πρασίνους. Καλώς ήλθατε, Υπουργέ. Χαίρομαι που είσαστε ο κύριος Γκρίλη και ο κύριος Γκρίλο. Ε, ίσως κάποια μέρα να έρθει και αυτός, κανείς δεν ξέρει, τέλος πάντων στις Βρυξέλλες, το αφεντικό σας, ε, θεωρείται ένα από τα πιο διακεκριμένα μέλη του Συμβουλίου και ίσως το μοναδικό μέλος που αντιτίθεται στην Άγγελα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ακούσω και την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας. Είχαμε εδώ πέρα τον Ζαν Πολ Γιούγκερ σήμερα και ξέρετε και τόσο δεν μας τα λόγια του. Και αναφέρθηκε στη γενική φύση του μείγματος πολιτικής που επιβάλλεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες από την αρχή της κρίσης και είναι Ανέφερα ότι δεν είναι βέβαιος ότι είναι το πιο σωστό μείγμα αυτό, γιατί μιλάμε συνεχώς για λιτότητα και κατανοούμε πλέον ότι ο μακροοικονομικός πώς δεν έχει νόημα αυτό και για την Γαλλία και για την Ιταλία και για το καθεξής και ότι τελικά πληρώνουν οι πιο αδύναμοι. Αυτό αφενός, αφετέρου είμαστε σε μια κατάσταση ασύμετρων σοκ, αλλά υπάρχουν, θεωρείται και ασύμετρες διορθώσεις ή θα πρέπει να είναι πιο συμμετρικές ε, οι διορθώσεις, αυτοί οι μηχανισμοί διόρθωσης, δηλαδή ότι θα πρέπει κάτι να κάνουν και οι χώρες με υψηλό πλεόνασμα. Να ακούσω λοιπόν την άποψή σας, όχι μόνο ως μέλος της Ιταλικής Κυβέρνησης, αλλά και ως μέλος του ΕΚΟΦΗΝ. Ευχαριστώ. Απάντηση. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να γίνει διάκριση. Όταν βρισκόμαστε εν το μέσο μιας ε, κρίσης, μέσα στην ομίχλη, ε, έχουμε ένα σχέδιο για το μέλλον της Ευρώπης. Νομίζω, ως οικονομολόγος, αν όχι ως εμπειρογνώμονας, ε, ούτε λόγιος, αλλά ως κάποιος που έχει σπουδάσει οικονομικά, ξέρουμε ότι τέτοιες περίοδοι ε, δημοσιονομικής προσαρμογής θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον κύκλο της ευρωπαϊκής οικονομίας μακροοικονομικά, τα μακροοικονομικά ουσιαστικά ε, εφευρέθηκαν για να απορροφήσουν τέτοιες κλειδονισμούς. Άρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλές από τις δημοσιονομικές προσαρμογές ε, που αναγκάζονται να κάνουν πολλές χώρες δεν ε, είναι εποφελής σε βραχή επίπεδο. Ωστόσο, όταν βρισκόμαστε μέσα στην ομίχλη, όπως ήμασταν πριν από κάποιους μήνες, μέχρι πριν από κάποιους μήνες, που μάλιστα ήταν πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση για πολλές χώρες, σε αυτή την περίπτωση το περιθώριο ελιγμού, το περιθώριο επιλογών για να επιδείξει κανεί μια χαλαρότητα σε ό,τι αφορά τι προσαρμογές αυτές δεν υπάρχει. Άρα σε κάποιες χώρες υπάρχει το ερωτηματικό. Θα συνεχίσουν αγορές να αγοράζουν τα ομόλογά μου, να με χρηματοδοτούν. Όταν το έχει και το θέτει αυτό μια χώρα σε ερώτημα, δεδομένης και της ε, κρίσης και της διάστασης τη κρίση θεωρώ, θεωρώ εγώ προσωπικά ότι χρειάζονται και ήταν αναπόφευκτες πολύ σκληρέ δημοσιονομικές προσαρμογές. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον, κατά πόσον θα σχεδιαστεί μια Ευρώπη χωρίς τους μηχανισμούς που αναφέρατε. Και αν αυτό θα είναι καλύτερος τρόπος απορρόφηση των κλειδονισμών, είτε με συμμετρικό είτε με ασύμμετρο τόπο. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν ε, περιπτώσεις που μπορεί όλη η περιοχή να ταλανιστεί από κρίση. Μετά από αυτά που συζητάνε οι ηγέτες στην Ευρώπη, φαίνεται ότι προσπαθούν να οικοδομήσουν έναν τρόπο για ένα καλύτερο σχεδιασμό της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των κρίσεων, για την απορρόφηση συμμετρικών και ασύμμετρων σοκ. Αλλά αυτό αποτελεί ασφαλώς μια διαδικασία. με διάφορα επίπεδα, με διάφορα βήματα και θα πρέπει να τεθούν και οι βάσεις. Και αυτή η βάση ήταν το Μουσουλμικό Σύμφωνο και ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Γιατί θεωρώ προκειμένου να υπάρχει ένας κοινός μηχανισμός ε, απορρόφησης κλειδονισμών θα πρέπει να είναι ένας μηχανισμός αυτός ο οποίος θα θετήθεται σε όλους. Άρα ήταν κάπως ατυχές ε, το, το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση με τόσο μικρή επιλογή σε ό,τι αφορά τις επιλογές κάθε χώρας δηλαδή. Νομίζω όμως ότι διδαχτήκαμε από αυτήν και ελπίζουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις αλλαγές αυτές, οι οποίες θεωρώ ότι είναι ευπρόσδεκτες. Μάλιστα, λέγει ο πρόεδρος, ο Μάρο, Μαουρό από την Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω. Για την Ιταλική κατάσταση. Αναφέρομαι σε ένα από τους δείχτες που τους μήνες μόλις ανέλαβε η υπηρεσιακή κυβέρνηση στην Ιταλία ακούστηκε πάρα πολύ. Ακόμα και στα κείμενα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφέρθηκε ως ε, ένας προβληματικός δείχτης για την Ιταλική πραγματικότητα. Δηλαδή η Ιταλική επίδοση ε, στην, αγορά των CDR. Μετά από 13 μήνες της κυβέρνησης Μόντι Άλλαξε τίποτα. Ε, άλλαξε ο τρόπος αντιμετώπισης του Ιταλικού χρέους. Εσείς μας μιλήσατε για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην επίδοση, επίδοσή μας σε αυτή την αγορά και ε, την πολιτική μας αξιοπιστία. Υπάρχει κάποια σχέση. Ευχαριστώ. Σίγουρα κάτι άλλαξε. Για να μην πω πολλά αρκεί να κοιτάξουμε και τα νούμερα. Τις πιο δύσκολες στιγμές της ε, κρίσης, αυτός έγινε ο πιο οικείος ε, ε, δείκτης, αυτό το credit default swaps, μαζί με τα spreads. Άλλαξε αυτός ο δείκτης, βελτιώθηκε και δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αγορές στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη γενικά. Βεβαίω τώρα επ' αυτού διαβάζουμε διάφορε γνώμε. Ορισμένοι λένε ότι αυτό οφείλεται στι προσπάθειε που έκαναν κάποιε χώρε ή στι προσπάθειε που έκανε η Ευρώπη ή στι προσπάθειε που έκανε άλλοι, στι προσπάθειε που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω ότι η ΕΚΤ έκανε μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την οικοδόμηση αυτών των μέτρων επίλυση τη κρίση της Ευρωζώνης. Δημιούργησε και εργαλεία και μηχανισμούς, αλλά και μια συνολική στρατηγική. Γιατί, όπως και εσείς ξέρετε, η ΕΚΤ σχεδίασε κάποια μέσα, κάποιες παρεμβάσεις και τα εξάρτησε από κάποιες προϋποθέσεις. Πολύ σημαντικές, κάτι την άποψή μου. να την άποψή μου, είναι απόλυτα Θετικέ αυτέ οι προποθέσει. Ο στόχος είναι να φτάσουμε σε αποτελέσματα όπου όλοι και τα θεσμικά όργανα και οι χώρες που πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα να συνεχίσουν να τα κάνουν. Αν δούμε χωριστά αυτές τις προσπάθειες που γίνονται και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΚΤ και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, αν τα πάρουμε μεμονωμένα, χωριστά κτλ., δεν θα αρκούσαν για να σταθεροποιήσουν τις αγορές. Κάθε συνιστός όμως ήταν αναγκαία για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Θα ήταν πολύ δύσκολο να σταθεροποιήσουμε τις αγορές, να σταθεροποιήσει τις αγορές μόνη της μια χώρα. Γιατί όπως είδατε, οι αγορές θεωρούσαν ότι υπήρχε ένας συστημικός κίνδυνος, ας το πούμε έτσι. είχαμε κάποιες, α, κάποιους κασανδρισμούς ας που θα μπορούσαν να επαληθευθούν μόνο και μόνο επειδή ακούγονταν. Επίσης, ήταν δύσκολο να σκεφτούμε ε, αξιόπιστες δημοσιονομικές πολιτικές χωρίς σημαντικές προσπάθειες, ορατές προσπάθειες σε, στο εσωτερικό, προσπάθειες μεταρρυθμιστικές στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Εμείς στην Ιταλία έχουμε βελτιώσει τα spread μας και αυτή η βελτίωση οφείλεται σε αυτό το συνδυασμό. Ο Πρωθυπουργό μας προσπάθησε να προωθήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθεροποίησης και μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας και παράλληλα να γίνει το ίδιο στην Ευρωζώνη. Δηλαδή και η κάθε μία χώρα της Ευρωζώνης να συνεισφέρει, αλλά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδίως. Κυρία Λούλιν από το Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, την ε, Πέμπτη είχαμε εδώ τον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος αποστασιοποιήθηκε από αυτή την πολιτική τη ε, λιτότητα. Αλλά πρόκειται βέβαια για το Eurogroup, το οποίο επί 8 χρόνια το προείδρευε και εκείνο το Eurogroup απίτησε αυτή την εξυγίανση των δημοσιονομικών όσον αφορά τα πιο χρεωμένα από τα κράτη-μέλη. Λέμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ πικρή, όμως πρέπει να καταλάβουμε κατά πόσο θα αποδώσουν καρπούς αυτές τις πολιτικές λιτότητες ή ου. Και ήδη μας είπε ότι είναι αντιπαραγωγικές, αλλά όμως έχουμε κάποιες ενδείξεις σε Ιταλία, Πορτογαλία, ακόμα και στην Ελλάδα. Που αυτές οι ενδείξεις μας οδηγούν στο να σκεφτούμε ότι υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι έχει οδηγήσει και σε κάποια ύφεση αυτή η πρωταδίσα πολιτική. Πιθανότητα την οποία την είχαμε υποτιμήσει. Άρα, τι να πιστέψουμε και ποιο να πιστέψουμε. Τι λέτε, τι πρεσβεύετε. Δύσκολη περίοδος. Θα συνεχιστεί, θα είναι μακρά ή ου. γιατί Έχουμε αυτό που είπε πρώτα του Eurogroup, που μια μεριά μας είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες πολιτικές ενώ η μεριά μας λέει ότι θα πρέπει να συρρυκνώσουμε το χρέος και το, και το, και το, και το, έλλειμμα. Μας λέει ότι για τα κάτι default Για τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σίγουρα πήραμε ένα χάπι πικρό, κάτι περισσότερο από πικρό χάπι μάλιστα. Βέβαια, το πόσο πικρό ήταν εξαρτάται και από τη χώρα. Κάποιες χώρες είχαν περιθώρια επιλογής. Μεγαλύτερα από άλλη. Εμείς δεν είχαμε πολλές επιλογές, πολλά περιθώρια στην Ιταλία. Είναι αδύνατο να δημιουργήσουμε μια στρατηγική ανάπτυξη αξιόπιστη χωρίς σταθερές χρηματαγορές. Είναι σαν να φτιάχνουμε ε, ένα σπίτι πάνω στην άμμο. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε ήταν να ξαναδώσουμε στις αγορές εμπιστοσύνη στη χώρα μας. Εμπιστοσύνη στην Ιταλία. Στο παρελθόν είμαστε μια χώρα οφειλέτης πρέπει, έπρεπε να δείξουμε στι αγορές ότι είμαστε αξιόπιστος ο Επομένως, όλα αυτά τα μέτρα σταθεροποίηση ήταν αναπόφευκτα, αλλά ήταν σημαντική και να γίνουν όλα αυτά με, μεγάλη ταχύτητα. Γιατί θεωρούσαμε ότι είναι σημαντική η ισοσκέληση του προπολογισμού μέσα στο 2013. Και εμείς και, το, και στο εξωτερικό ε, θεωρούσαμε ότι αυτό είναι αποφασιστικό μήνυμα που θα στέλναμε ως Ιταλία στις αγορές για να αποκτήσουμε την αξιοπιστία μας. Φυσικά η λιτότητα δεν είναι αυτός σκοπός, είναι μέσο για να οικοδομήσουμε εν συνεχεία την ανάπτυξη. Ο κύριος Γιούνκερ νομίζω μίλησε για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ανάπτυξη που ξεπερνάει την απλή πολιτική λιτότητα. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η συζήτηση, αυτό το επιχείρημα συζητήθηκε στην Ευρώπη. Θα θυμάστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Ορισμένοι το θυμούνται μόνο για τα επιχειρήματα ε, λιτότητας. Αλλά όχι, εκεί αρχίσαμε να μιλάμε και για επενδύσεις. Για κοινέ επενδύσεις, ε, ευρωπαϊκή προσπάθεια επενδύσεων με πιο αυξημένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζος ε, Επενδύσεων. Έχουμε λοιπόν δύο παράλληλα πράγματα που προχωρούν παράλληλα. Δυστυχώς στην Ευρώπη ε, μόνο σε ορισμένες αγορές είδαμε τη σταθερότητα των αγορών, ε, όπως στην Ιταλία. Ε, εμφανίστηκε πρώτα αυτό το σκέλος, χωρίς το επόμενο το συνοδευτικό σκέλος. αλγευρικά. Είναι εύκολο να φανταστούμε μια ισοσκέληση των λογαριασμών, αλλά είναι πιο δύσκολο να σκεφτούμε με ποιον τρόπο θα τροφοδοτήσουμε εκ νέου την ατμομηχανή της ανάπτυξης. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε και μεμονωμένα και συλλογικά ως Ευρώπη. Και τώρα η κυρία Κλέμα για τους σοσιαλιστές από τη Σλοβενία. Γεια σας, θα, μιλήσω στα αγγλικά. Στους τελευταίους μήνες υπολόγισαν κάποιες ερευνές ότι λόγω της φοροδιαφυγής ένα τρισεκατομμύριο χάνει η Ευρώπη κάθε χρόνο σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρήμα και θεωρώ ότι αυτοί οι σκανδαλώδεις ε, νόμοι στην εθνική νομοθεσία αποτελούν μία απειλή για τα κοινωνικά μοντέλα σε ό,τι αφορά και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά την καλή ε, λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Αυτή η απώλεια εσόδων εξακολουθεί να απειλεί πολλά κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καιρούς κρίσης Προφανώ θα έπρεπε να έχει θέσει αυτό το θέμα στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Και αυτό οδηγεί σε μείωση των ε, δαπανών για την καταπολέμηση της ενεργείας και της οικονομικής κρίσης. Είμαι εισηγήτρια σε μια σχετική έκθεση για τη φοροδιαφυγή. Θα καλέσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, να αναλάβουν δράση για να καταστρώσουν και να καταρτήσουν μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική και θεωρώ ότι από κοινού θα μπορέσουμε να μειώσουμε κατά 50% τα κενά αυτά στη φορολογία μέχρι το 2020 και επειδή η Ιταλία είναι από τα κράτη-μέλη με το υψηλότερο ποσοστό σκιώδους οικονομίας, μαύρης οικονομίας, με τεράστια ποσοστά λοιπόν τέτοια, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα εθνικά μέτρα τα οποία έχετε εισαγάγει προς το σκοπό αυτό και τι πρέπει να γίνει ακόμα, γιατί έχουμε ακούσει πολλά σχετικά τους τελευταίους μήνες από την Ιταλία και επίσης να ακούσουμε την άποψή σας και τη θέση σας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. η φοροδιαφυγή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Κοινό σε όλες τις χώρες. Αλλά είναι πολύ πιο οξύ σε ορισμένε χώρες. Και δυστυχώς η Ιταλία είναι διαβόητη γιατί έχουμε ένα επίπεδο φοροδιαφυγής πολύ πιο ψηλό από το μεσόωρο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που η κυβέρνησή μας ε, εντόπισε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τη στιγμή λοιπόν που κάναμε την πρώτη προσπάθεια δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και σταθεροποίησης, μία... κάναμε ιδιαίτερη προσπάθεια για να τροποποιήσουμε τη στάση μας απέναντι στη φοροδιαφυγή. Καταρχάς χάνουμε πόρους. Αλλά υπάρχει και θέμα δικαιοσύνης φορολογικής δικαιοσύνης. Πρέπει να δούμε όμως και την έλλειψη πόρων που χάνουμε ε, και εξαιτία αυτού δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ε, κοινωνικά προγράμματα. Επομένως υπάρχει ε, μια διπλή αδικία στην φοροδιαφυγή. Υπάρχει και μια τρίτη αδικία του level playing field, της ισοτιμίας μεταξύ διαφόρων επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Γιατί αν υπάρχουν διάφορε, διάφορες που ανταγωνίζονται στην αγορά. Κάποιες φοροδιαφεύγουν. Αυτές που φοροδιαφεύγουν έχουν α, προφανώς ένα πλεονέκτημα που είναι φυσικά αθέμητο, που είναι παράνομο. Ε, για οικονομικούς λοιπόν και κοινωνικούς λόγους πρέπει να καταπολεμήσουμε ε, το, τη φοροδιαφυγή. Έχουμε εισαγάγει πολλά μέτρα που σκοπό έχουν να ενισχύσουν την ε, ικανότητα των φορολογικών μας αρχών της εφορίας μας να γνωρίζει το πρόβλημα, να ιχνηλατεί και τις ε, συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών μας. Αυτό, αυτή η προσπάθεια δίνει καλά αποτελέσματα. Φυσικά πρέπει να αλλάξουμε και νοτροπία. Όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι φορολογικές αρχές. Υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης σήμερα, πληροφόρησης. Θα πρέπει λοιπόν και οι φορολογικές αρχές να υποφεληθούν από αυτή τη δυνατότητα. Είμαστε στην πρώτη χρονιά εφαρμογής. Την πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε μάλλον είχα, με μια μεγάλη ε, οικονομική αδυναμία. Επομένως είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα των μέτρων. Επιπλέον, σε, στιγμή, σε στιγμές οικονομικών δυσκολιών, αυτή η αλλαγή νοοτροπίας και από τους πολίτες και από τις αρχές είναι πολύ σημαντική. Μια και μιλάτε τόσο καλά τα Ιταλικά, φαντάζομαι θα μπορείτε να διαβάσετε και τις Ιταλικές εφημερίδες και θα βλέπετε ότι υπάρχουν πολύ έντονα επιχειρήματα για να, προσπαθει... να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα έτσι διάχυτο κλίμα φόβου αβάς όταν δεν χρειάζεται. Θα πρέπει να εξηγήσουμε πολύ σωστά όλες αυτές τις αλλαγές, να τις δικαιολογήσουμε για να διασκεδάσουμε τους όποιους φόβους. Ευχαριστώ πολύ. Να, μία λίστα ήταν. να τα δει κανεί σοβαρά και να φυλακίσει κάποιον που έχει τέτοια ολιστήματα όπως τον πρώην Πρωθυπουργό σας. Σαμπίν Κούτας τώρα, σοσιαλιστής από τη Ρουμανία. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ πρώτα πρώτα που ήρθατε να μας επισκεφτείτε. Χωρίσατε σε δύο μέρη την ομιλία σα, πρώτα για την Ευρώπη και εδώ για την Ιταλία. Οπότε και εγώ να σα πω αντίστοιχα τι ερωτήσει μου, μια ερώτηση για την Ευρώπη και μία για την Ιταλία. Τώρα, όσον αφορά την Ευρώπη, όπω ακούσατε προέρχομαι από την Ρουμανία, που ακόμα δεν έχουμε μπει στην Ευρωζώνη. Εσεί είστε από την Ιταλία που είστε στην Ευρωζώνη και γι' αυτό σα ερωτώ, ποια είναι η γνώμη σα για αυτή την καινούργια ιδέα που έχει παρουσιαστεί για την Ευρώπη δύο ταχυτήτων μάλλον θα ξέρετε ότι έχει αναφερθεί το να έχουμε και δύο κοινοβούλια, τον για την Ευρωζώνη και ένα για την υπόλοιπη Ένωση. Είχαμε και τις συζητήσεις για τις τράπεζες και είπαμε πίσω ότι σε σχέση με την τραπεζική υποπτία, τραπεζική ένωση έχουν πιο πολλά δικαιώματα οι χώρες της Ευρωζώνης. Παρά το ότι πλέον ότι οι τράπεζες βρίσκονται παντού και στη Δε Ρουμανία το 1% της αγοράς το έχουν καταλάβει οι τράπεζες χωρών της Ευρωζώνης. Για πέστε μας πώς τα βλέπετε εσείς για αυτή την ιδέα που κυκλοφορεί για το... Και ποιο, και ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης αν το πάμε έτσι. Δεύτερον. Για πέστε μου για την Ιταλία. Μας είπατε τα μέτρα της διαφθοράς, η περισσότερη διαφάνεια για να ελκύσετε επενδύσεις. Εγώ απορώ αυτά που διαβάζω για αυτό το νέο φόρο. Ε, αυτό το, το, το δημοτικό φόρο. Αυτός ο νέος φόρος, λοιπόν, πώς θα εισπράττεται. λέτε ότι αυτός ο φόρος θα είναι τώρα κατά αποκοπή ίδιος για όλους. Τι λέτε. Τι θα γίνει όταν λοιπόν επιβληθεί η κυβέρνησή σας. Ο Υπουργός. Σας ευχαριστώ. Για την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. εγώ Στην βαθιά στην Ευρώπη και στο ευρώ. Ε, όμως δεν υπάρχει αυτό με τους πιλότους. Μόλις βγούμε από το τούνελ της κρίσης και έχουμε μπορέσει να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις στη, για τη διακυβέρνηση, να βρούμε μέτρα για πρόληψη των κρίσεων, ε, τότε η Ευρωζώνη και η Ευρώπη θα ταυτίζονται άντε με μια εξαίρεση. Αλλά αυτά τα ορίζει η συνθήκη. Άρα κανείς θα πρέπει να έχει τέτοιου είδους πεποίθηση, όχι απλώς να ελπίζει. Και επομένως Ευρώπη και Ευρωζώνη συγκλίνουν. Θα πρέπει υπάρχει άλλο σεβασμός για τις ελευθερίες του ε, εκάστου. Άρα αντίστοιχα σεβασμός και για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Και έτσι οι αποφάσεις της Ευρωζώνης να μην θέτουν να την ελευθερία αυτή. Η ελευθερία μπέσω δώσει μέσα στο κοινό πλαίσιο. Από την άλλη μεριά θα πρέπει υπόψη τις ε, ανάγκες των μελών της Ευρωζώνης, μια που οι χώρες αυτές είναι προσδεδεμένοι μια στην άλλη και θα πρέπει επομένω να τις προχωρήσουμε μέσα σε ένα στοιχειώδες, λογικό, χρονικό πλαίσιο. Αυτά μας το πρέπει να εξορροπήσουμε. δύσκολο έργο και περίπλοκο. Εγώ όχι, εγώ θεωρώ ότι το να κατατιμήσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είναι η ιδιώδης λύση. Θα πρέπει να γιατί ως αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου το πρόβλημα του. Θα πρέπει να έχουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε δόκιμα ή όχι ελευθερία, αλλά για την άλλη μεριά να μπορέσουμε να έχουμε το περιθώριο για κάποιε κοινέ αποφάσει που θα πρέπει να ληφθούν για τα μέλη τη Ευρωζώνη και καμιά φορά με τρόπο κατεπήγοντο τρόσον αφορά την Ιταλία και αυτό τον φόρο του περιουσίας το πνεύμα του φόρου αυτού ήταν αυτό να αφορά κάθε είδους εμπράγμα του δικαιώματος. Έχουμε ράβει ξύλωνα πέραν τις πρώτες κατοικίες πέρασε τώρα ένας χρόνος οπότε τώρα ακριβώ κάθε είδους ακίνητο φορολογείται λιγότερο για την πρώτη κατοικία, περισσότερο γιατί έχει κανείς πέραν αυτής. Βεβαίως. έχουν ψηλό το ίδιο κατοίκη στην Ιταλία, όπως ξέρετε. 80% περίπου των Ιταλών είναι κύριοι τουλάχιστον ενός ακινήτου. Αυτά πρέπει να επιβληθεί αυτή είναι η αφορολογία η οποία θα επιβληθεί σε όλους τους Ιταλούς. Ποτέ φυσικά δεν είναι καλοδεχούμενη μια φορολογία. Τι, να σας πει εκείνη η γνώμη. Θέλετε να κατέβουν στους δρόμους και να πανηγυρίζουν. Παρ' όλα αυτά. Εάν κάνετε μια συγκριτική μελέτη, περισσότερες χώρες έχουν ένα τέτοιο φόρο που επιβάλλεται επί κάθε είδους ακινήτου. Αυτά. Τώρα, το αν είναι αναλογικός ένας φόρος ή όχι, αλλά γενικά είναι καλό να είναι ένας φόρος αναλογικός. Αλλά ούτε αυτό είναι αυτό να ρίξετε μια ματιά τι γίνεται σε όλες τις χώρες γιατί όπως ο προηγουμένος με αυτό το φόρο εξασφαλίζουμε έσοδα για τις τοπικές αρχές. Εκεί είμαστε πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον ισχύει αναλογικότητα, κάτι το οποίο δεν είναι επίσης πάρα πολύ απλό και ούτε αυτό ισχύει στις περισσότερες χώρες ακριβώς γιατί πρόκειται για πηγή εσόδων για τις τοπικές αρχές και επίσης Πάρα πολλέ φορέ, τα ακίνητα δεν ανήκουν σε κάποιο φυσικό πρόσωπο, ανήκουν σε κάποιο είδου εταιρείε. Άρα ούτε εκεί είναι απλό το να θεωρήσουμε ότι ισχύει, να δούμε πώ θα εφαρμόσουμε το στην αναλογικό του πρόεδρος. Για βάλτε τα λευκά σας να σα ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι φιλελεύθερος Γερμανός ευρωβουλευτή, ο κύριο Μπερσάνη. Αν σα τα πω στα γερμανικά. Κύριος Βερσάνη, ο οποίος ε, είναι υποψήφιος ε, πρωθυπουργός, ε, έχει δηλώσει ότι αν ε, βγει πρωθυπουργός θα ξαναδιαπραγματευτεί μία σειρά συμβάσεων που έχουν συναυθεί τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες γιατί θεωρεί ότι δεν συμφωνεί με αρκετούς όρους και θέλει να τους επαναδιαπραγματευτεί. Και έτσι θα βρισκόμασταν στη σε κατάσταση. Το σύμφωνο σταθερότητας ε, και δεν έγινε σεβαστό και αυτό μα θεωρείται ότι είναι προεκλογική στρατηγική ή ότι πρόκειται να το κάνει πραγματικά ο κύριος Βερσάνη τώρα σε ό,τι αφορά ε, τη σχέση του ευρώ σε σχέση με άλλα νομίσματα στον κόσμο. Είναι καθοδική η τάση του ευρώ η τράπεζα της Ιαπωνίας ε, και άλλες ε, τράπεζες το σπρώχνουν προς τα κάτω το ευρώ. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνουν και οι Αμερικανοί με την πάροδο του χρόνου για να βελτιώσουν ε, την ανταγωνιστικότητά τους με το δικό τους νόμισμα. Τι θεωρείτε ότι είναι κρίσιμο σε ό,τι αφορά την συναλλαγματική συντομία μεταξύ ευρώ και δολαρίου για να αποφύγουμε αυτό το μάτσα, αν θέλετε, μεταξύ συνταγματικών ισοτιμιών. Πρόεδρε, εσείς ο ίδιος είπατε ότι είμαστε κυβέρνηση εμπειρογνωμόνων, κυβέρνηση γραφειοκρατών, υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν είμαστε πολύ καλοί στη συζήτηση των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων. Τα κόμματα τώρα ξεκινάνε την προσπάθειά τους για τις εκλογές. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω σε αυτή τη φάση αν αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις τακτικής ή όχι. Κάποια στοιχεία θέλω να δώσω. Η Ιταλία και το Ιταλικό Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα τα οποία υποστήριξαν την κυβέρνηση Μόντι όχι μόνο ενέκριναν το περιεχόμενο του Fiscal Compact, του Δημοσιονομικού Συμφώνου, αλλά το πήραμε πολύ στα σοβαρά. Είμαστε μία από τις χώρες, μία από τις λίγες χώρες, ακόμα και σήμερα νομίζω, που έχουν ήδη εισαγάγει στο Σύνταγμά τους, όπως είπα πριν, ένα βασικό στοιχείο της δημοσιονομικής πειθαρχία που υπήρχε στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και που είναι η ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Και το Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο ε, πέρασε τον ενισχυμένο νομοσχέδιο, όπου αναφέρουμε με λεπτομέρεια πώς αυτό το επιτυγχάνουμε κάθε χρόνο. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ να σας καθησυχάσω από αυτήν την άποψη ότι τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ε, αυστηρότητα των δημοσίων λογαριασμών και την ε, ισορροπία του προϋπολογισμού την έχουμε γράψει στο σύνταγμά μας. Ε, είμαστε βαθιά Πεπισμένη γι' αυτό και για να περάσει αυτή η συνταγματική αλλαγή υποστηρίχθηκε από μια ευρία πλειοψηφία. Και αποτελεί τώρα αυτό τμήμα του θεσμικού μας πλαισίου, του συνταγματικού μας πλαισίου. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να το αναθεωρήσουμε αυτό. Γιατί χρειάστηκε μια ευρύτατη πλειοψηφία που ένα κανονικό κοινοβούλιο σε κανονικές συνθήκες δεν επιτυχάνει. Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστική υποτίμηση, βλέπουμε ότι η Ιταλική θέση και η Ευρωπαϊκή θέση πάντα ήταν, ήταν πάντα αντίθετη στην χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών για εμπορικούς λόγους. Δεν είμαστε υπερπολιτικών αλλαγή της ισοτιμίας, η τρέμβαση στις αγορές συναλλαγματικών ισοτιμιών. Έχω αρνητική στάση στο να χρησιμοποιούμε συναλλαγματικές ε, ισοτιμίες για εμπορικούς σκοπούς ο τρόπος που οικοδομήθηκε μάλιστα το ευρώ και θα θυμάστε την εμπειρία της χώρας σας, πρόεδρε, της Γερμανίας. Μια χώρας με μεγάλη επιτυχία στις εξαγωγές. Ε, η Γερμανία είναι ε, πιστικός ανταγωνιστής στις ε, παγκόσμιες αγορές χωρίς να χρησιμοποιεί τη συναλλαγματική ισοτιμία. Μπορεί να είναι δηλαδή να έχει κανείς ισχυρό νόμισμα, ισχυρή ισοτιμία, ισχυρή οικονομία, χωρίς να παίζει εκεί. Γιατί μια τέτοια πολιτική μπορεί βραχυπρόθεσμα να αποδώσει, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι αρνητική κατά την άποψή μου. οι επιχειρήσεις μας ε, και οι, κυρίως οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν αρνητική στάση για αυτή τη θέση μας βέβαια. Αλλά εμείς πάντα λέμε ότι τέτοιες πολιτικές δεν είναι συμβατές με την ιδέα της ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύριος από τους συντηρητικούς και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα λιτότητα τη ε, απερχόμενη Ιταλική κυβέρνηση ουσιαστικά εκφράστηκε σε υψηλότερη φορολόγηση και στο World Sleep Journal πέρσι ο κύριο Δράγκη ε, το ανέφερε αυτό ω κακή εξυγίανση με αντίθετη την καλή εξυγίανση με χαμηλή φορολόγηση. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα περιοριστούν οι υπερβολικές δαπάνες ε, της κυβέρνησης. Ε, ο Βόλφαρ Μουνχιάου υποδεικνύει σήμερα σε μια συνέντευξη ότι οι μεταρρυθμίσεις του κυρίου Μόντι θα είναι ασήμαντες μακροοικονομικός πώς. Πώς σχολιάζεται και τα σχόλια του κυρίου Δράκη και του κυρίου Μουνχιάου και ποιε είναι οι τριφωτικέ ε, μεταρρυθμίσει που χρειάζονται για να υπάρξει εκ νέου ανάπτυξη στην Ιταλία. to... Να σα αναφέρω ποια είναι τα περιστατικά και όχι ποια είναι η άποψή μου. Τα γεγονότα. Η γνώμη μου όντω είναι ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε από την αρχή της κυβέρνησής μας η ανάγκη εξυγίανσης των δημοσιονομικών ήταν τέτοια και έπρεπε να ολοκληρωθεί σε τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο της φορολόγησης περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε και εμείς οι ίδιοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε σε αυτό. Δεν, δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει γίνει το αντίθετο και να σας πω ότι ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι να περιοριστούν τα, οι δημόσιες δαπάνες για να, να μειωθεί ο δημόσιος τομέας και στην Ιταλία σήμερα τι κατοχυρώνει το Σύνταγμα όταν ε, οι κυβερνητικές διαπάνες είναι ίσες με το φορολογικά έσοδα, αν θέλει κανείς να περιορίσει τη φορολογία θα πρέπει να μεταρρυθμίσει ριζικά και τις ε, δημόσιες δαπάνες. Αυτό δεν το ξεχάσαμε. Κάναμε δύο ασκήσεις για τη μεταρρύθμιση των δαπανών. Ε, περιορισμό των κυβερνητικών προγραμμάτων. Στον ένα χρόνο που είχε στη διάθεσή της η κυβέρνηση αυτή Και η άποψή μου και η άποψη του Προέδρου θεωρώ είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί και το φορολογικό βάρος. Και όταν αυξάνουμε την φορολογία προσπαθούμε να το κάνουμε με έξυπνο τρόπο, να απομακρυνθούμε από τη φορολογία εισοδήματο, για παράδειγμα, και να κινηθούμε προς την φορολογία των ακινήτων. Αλλά γενικά η συνολική φορολόγηση θα πρέπει να μειωθεί, θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί όπως είπατε και το ζήτημα των δαπανών, των δημοσίων δαπανών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό φυσικά είναι και θέμα επιλογών. Και είναι δύσκολες ε, οι επιλογές αυτές. Είναι δύσκολο να αυξήσει κανείς ε, τη φορολογία, αλλά είναι και δύσκολο να συρρυκνώσει τον δημόσιο τομέα. Υπάρχουν πολλές δημόσιες ε, κοινοφελείς υπηρεσίες κτλ. κτλ. Είναι σαφής λοιπόν η ανάγκη για πολιτική καθοδήγηση στη διαδικασία αυτή. Το σχόλιο του Πρόεδρου Ντράκη τώρα. Ξέρετε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν χώρες όπου οι δημόσιες δαπάνες και η φορολογία δεν μειώνονται, αλλά αντιθέτως αυξάνονται. Αλλά αυτό εξαρτάται και από τις κοινωνικές συμβάσεις στην κάθε χώρα. Θεωρώ ότι στη δική μου χώρα η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να μειωθούν οι φόροι. Και άρα το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τις δημόσιες δαπάνες. Ο κ. Μόντσαου, σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα, σέβομαι αυτά που γράφουν οι Financial Times και σίγουρα αποτελούν μέρος του διαλόγου. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, και όσα αποφάνθηκε για το κατά πόσο ήταν συνεπή και συνεκτικά τα μέτρα που εφαρμόσαμε και θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχει μια τέτοια συνοχή. uh, our... Ο πρόεδρος Κλίντς. Η συνάδελφος Περβάν Περέες ζήτησε το λόγο, αλλά δυστυχώς ε, βρίσκεται σε άλλη επιτροπή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ο Τζόνι Πιτέλα ζήτησε το λόγο ανταυτής. Παίρνω ξανά το λόγο για μια διευκρίνηση. Ο πρόεδρος Κλίνς, που είναι αξιοσέβαστο πρόσωπο, όχι μόνο κάτι γνώμη μου, αλλά και κατά γνώμη όλης της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Σίγουρα είναι, οδηγήθηκε σε λάθος από παραπληροφόρηση. Ο Λουίτζι Μπερσάνη, που είναι ο αρχηγός του κόμματός μου και της κεντροαριστεράς στην Ιταλία, γράφει λέξη προς λέξη δεν θέλω να επαναδιαπραγματευτώ το φορολογικό σύμφωνο, ούτε καμία από τις συμφωνίες που επιτύχαμε το τελευταίο χρόνο. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε προς τα εμπρός για την ανάπτυξη. Και επομένω να προωθήσουμε πολιτικές που συνδυάζουν την λιτότητα, που δεν την αμφισβητεί ο Μπερσάνη, με την ανάγκη να αυξήσουμε τις δημόσιες επενδύσεις και την απασχόληση. Ισχύει λοιπόν το σύμφωνο ο Μπερσάνη θέλει να διατηρηθούν όλα τα σύμφωνα τα οποία έχουμε επιτύχει στην Ευρώπη. Θέλουμε παράλληλα να υπάρχει όμως και μία, ναι, παράλληλα με τη λιτότητα να υπάρχει και μία πιο έντονη πολιτική υπέρ της ανάπτυξης και υπέρ της απασχόλησης. Ευχαριστώ Τζάνι για τις διευκρινήσεις. Τόσο το καλύτερο. Έτερος, Ζων Πόλου σύντομα θέμα, γιατί έχουμε όλες λεπτά, κύριε Υπουργέ. Σα ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από την αρχή που αρχίσατε και ακούγοντά σα όσον αφορά τις, ε, τη μεταρρύθμιση, την ε, δημοσιομική πολιτική, όσον αφορά τα, τα μέτρα τα οποία λάβουμε. Αναρωτιέμαι, τι θα πει κυβέρνηση τεχνοκρατών, τι εστί. Δύσκολη ερώτηση. Η διαφορά ίσως είναι ότι οι τεχνοκράτες δεν ανήκουν σε πολιτικές ομάδες, ε, σε πολιτικά κόμματα, αλλά δεν προέρχονται από το κοινοβούλιο, αλλά από την κοινωνία των πολιτών. Και όταν όμως μια κυβέρνηση αναλαμβάνει, όποια και αν είναι αυτή η κυβέρνηση, προβαίνει σε πολιτικές ενέργειες. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Η δική, η μας κυβέρνηση ήταν η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ε, κυβέρνηση εμπειρογνωμόνων, γιατί τα περισσότερα μέλη της κυβέρνησης αυτής δεν ανήκαν σε πολιτικά κόμματα, δεν ήταν πολιτικοί, δηλαδή δεν, ανήκαν στο, δεν το κοινοβούλιο. Αλλά μέσω της δράσης τους προβήκαν σε πολιτικές ενέργειες όταν έφτασαν ενώπιον του κοινοβουλίου και πρότειναν διάφορα πράγματα. Επομένω, μπορούμε να πούμε ότι πολιτική και τεχνική, ε, δηλαδή εμπειρογνωμοσύνη, είναι δύο πράγματα αλληλένδετα. Είναι πολιτικο-φιλοσοφικό το ερώτημά σα. Είναι η καλύτερη απάντηση που μπορώ να δώσω. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη ευχαρίστηση αλλά και τιμή το που ήρθατε να πέρασετε την ώρα μαζί μα. Ξέρουμε τώρα θα πρέπει να πάτε να συναντήσετε του ε, συναδέλφου σα για τη συνάντηση της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και πάλι. Έχουμε σημαντική εναλλαγή προέδρων σήμερα. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Ε, είναι τρεις σημαντικές εκθέσεις ε, που τις ετοίμασε ο Βέρνερ. Έχεις το λόγο. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ηλικία, είναι θέμα σοφία το γεγονό ότι μπορεί κανεί να προεδρεύει. Και άρα να ευχαριστήσω του ε, δύο συναδέλφου που παρά τι δύσκολε καιρικέ συνθήκε κατάφεραν να αντικαταστήσουν του προέδρου. Εγώ κατέθεσα γνωμοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις, όχι εκθέσεις, γιατί αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Ελέγχου Προεπιλογισμού Και άρα, στις 10 Ιανουαρίου του 2013, οι απαλλαγές αυτές οι τρεις για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων έλαβε χώρα λοιπόν μια ακρόαση κατά την οποία προσήλθαν ε, οι διευθυντές και τοποθετήθηκαν και δικαίως ε, έγινε αυτή η ακρόαση. Να σας πω ότι και στις τρεις περιπτώσεις ε, οι αρχές αυτές δημιουργήθηκαν για την ε, πιο αυστηρή διαμόρφωση των σχετικών διατάξεων και είναι το πρώτο έτος ουσιαστικά που χορηγείται απαλλαγές. Δεν είναι αυτόνομοι οι οργανισμοί αυτές οι αρχές, είναι κοινοτικές ε, αρχές ευρωπαϊκές και των κρατών ομαλών. Και εδώ ξεκινά το πρώτο πρόβλημα. Πώς θα διασφαλιστεί η χρηματοδότηση. ...60% κράτη-μέλη, 40% ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός. Αυτό ισχύει και για τις τρεις ε, αρχές και αυτό προκαλεί προβλήματα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι εθνικοί ελεγκτές έχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Το γεγονός ότι τα μέσα που δεν δαπανώνται επανεισραίουν. Το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση για άσκηση επιρροής. Και αυτό οδηγεί στο ερώτημα εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία που θέλει το Κοινοβούλιο. Το θέμα του πώς ε, η μείωση του προπολογισμού έχει επιπτώσεις ε, στην χρηματοδότηση, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Όλα αυτά, λοιπόν, ε, καταδεικνύουν ότι δεν είναι σαφής το δικό δόμημα των τριών αυτών αρχών. Και αυτό καταδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί κανείς να συμφωνήσει για μια τραπεζική ένωση ενώ λείπουν τα βασικά θεμέλια. Τα αποτελέσματα και τα πορίσματα των ακροάσεων των τριών διευθυντών τα διάβασα με μεγάλη προσοχή και τα αξιολόγησα από πλευράς ε, Επιτροπής ε, προεπολογισμού συστάθηκε να χορηγηθεί η απαλλαγή και να τεθούν ως προβλήματα τα θέματα του προσωπικού και τα χρηματοδότηση 60-40. Αυτά γενικά ως παρατηρήσεις. Να ξεκινήσω τώρα από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Το πλέον μιας γνωμοδότησης έχουμε θέματα και περιορισμού της ε, έκτασης της γνωμοδότησης. Καλούμαστε να τοποθετηθούμε. Να σας πω ότι στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταδεικνύει ότι υπάρχει αξιοπιστία δεν είναι ίσως το βέλτιστο αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα καλό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ε, δικαιοσύνη και την έλλειψη ατασταλιών. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τραπεζών, ε, δαπανήθηκαν τμήμα μόνο των της χρηματοδότησης και κάποιοι από τις στόχοι δεν επιτάχθηκαν. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, γιατί οι τρεις αρχές αυτές ξεκίνησαν από το μηδέν. Οι ανάλογες ε, αρχές σε εθνικό επίπεδο όλων των κρατών μελών έχουν 53.000 υπαλλήλους και καταλαβαίνετε ότι αναγκάστηκαν να αναλάβουν αρμοδιότητες οι οποίες ήταν κατά τα συμφερόντων των κρατών μελών. Και χωρίς κατάλληλη χρηματοδότηση κλήθηκαν να τις ε, επιτελέσουν τις λειτουργίες αυτές. Το ελεκτικό συνέδριο βρήκε τρία αδύναμα στοιχεία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Τραπεζών. Χρειάζεται ασφαλώς ε, να διασφαλιστεί η γρήγορη επαλήθευση όλων αυτών, γιατί ε, υποβάλλει προτάσεις για όλες τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις δικασίες προμηθειών και στις τρεις περιπτώσεις δεν συνάδουν απόλυτα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον γενικό προεπιλογισμό της Ένωσης και σε μία περίπτωση τηρήθηκαν εθνικές ε, διαδικασίες προμηθειών εγώ το ξέρω, αν και δεν αναφέρεται στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, ότι σε μία περίπτωση έγινε μία παράταση σύμβασης χωρίς να γίνει εκ νέου εξέταση των διαδικασιών προμηθειών. Και έτσι προέκυψαν πάρα πολλοί υψηλά ποσά μισθώσεων, πολύ πιο υψηλά από την τιμή της αγοράς. Επίσης, η αξιοπιστία και η διαφάνεια, η διαφάνεια και οι μισθοί τέθηκαν ως θέμα από το ελεγκτικό συνέδριο. Η αρχή εξέτασε τις περιπτώσεις αυτές και δήλωσε ότι πρόκειται να τις ρυθμίσει στο σημείο 7 παρακαλώ το ελεκτικό συνέδριο να ελεγξει επλεπτομερώς το 2013 τις δεσμεύσεις της αρχής για αποκατάσταση των λήψεων. Άρα, τους δίνουμε και κατανοούμε πόσο δύσκολη είναι η κατάστασή τους επειδή είναι και μια νέα αρχή, αλλά υπάρχει ανάγκη να τηρούνται οι ευρωπαϊκές διατάξεις, γιατί δεν δεν μπορούμε να κάνουμε έκπτωση. Αυτά για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Να συνεχίσω. Πολύ ωραία. Επόμενο. Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, η ΕΣΜΑ. Στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών παρέστη ο κύριος Βάκας, στην ε, ακρόαση, στην ε, ΕΣΜΑ ο κύριος Ρος, ο Βέρνερ Ρος. Παρόμοια είναι η κατάσταση, αλλά με κάποιες διαφορές σε ό,τι αφορά τα μεμονωμένα στοιχεία. Συνολικά το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι υπάρχει μια ακριβωτή και εικόνα και είναι κάπως πιο θετική η έκθεση από τη για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, αλλά και εδώ υπάρχουν χαμηλά ποσοστά εκτέλεση του προπολογισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν δυσκολίες κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση του προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τις ε, νομικές υποχρεώσεις. Δεν είναι δυνατόν να αναλυφθούν πριν από τον καθορισμό των ανλήψεων υποχρεώσεων. Πιστώσεις πληρωμών 200.000 ευρώ που δεν, στις οποίες δεν αντιστοιχούν καμία νομική υποχρέωση θα πρέπει να κυριευθούν και στο μέλλον να αποφευχθούν. Επίσης το Ελεκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η ΕΣΜΑ πρέπει να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν διατάξει εφαρμογή που αφορούν το καταστατικό των υπαλλήλων και μια διοργανική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία πολέμηση τη Απάτη. Δεν ξέρω πού ακριβώ εστιάζονται αυτά τα προβλήματα με την ΟΛΑΦ, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία πολέμηση τη Απάτη. Το ανέφερε αυτό το ηλεκτρικό συνέδριο. Γιατί δεν θεωρώ ότι η Όλαφ, ε, ε, ο σκοπό, η, μάλλον η δημιουργία της Όλαφ είχε σκοπό να δημιουργήσει μια αρχή με δικαστικές εξουσίες. Αυτό το κοιτάξω λοιπόν αυτό το σημείο, το αναφέρω απλά επειδή το ανέφερε και το ηλεκτρικό συνέδριο. Και εδώ αναφέρουμε ότι θα πρέπει να καλυφθούν το δυνατόν οι ελλείψεις της διαφάνειας των διαδικασιών πρόσληψης και του ορισμού και θα πρέπει να οριστεί μια εξεταστική επιτροπή ω νόμιμη διάδοχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών και των Αξιών. Επειδή υπάρχει αυτό ο προκάτοχο τη ΕΣΜΑ, Το θέμα τίθεται λοιπόν και για τα νίκια στο Λονδίνο. Ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό και εδώ στο 8 της γνωμοδότησης παρακαλώ το ελεκτικό συνέδριο να εξετάσει λεπτομερώς το 2013 τις ποικίλε ελλείψεις που εντοπίστηκαν. Η τρίτη τώρα αρχή. Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Και εδώ ε, εκφράζεται από δοκιμα... επιδοκιμασία για την ε, αξιοπιστή των και την ομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων. Δυσκολίες ε, στη φάση δημιουργίας. Οι δαπάνες λειτουργίες της υπηρεσίας ήταν πάρα πολύ χαμηλές και δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούσαν τον εξοπλισμό της αρχής. Το λογιστικό σύστημα, το λογιστικό σύστημα θα πρέπει να επικυρεθεί το συντομότερο δυνατόν και εγκύρος. Επίση, είναι απόλυτα αναγκαία οι των προμηθειών, είναι απόλυτα συμβατέ με τη διατάξει του δημοσιονομικού κανονισμού, τα κριτήρια ανάθεση να ορίζονται εκ των προτέρων, οι συμβάσει να παρουσιάζονται σε γραπτή μορφή και να τηρούνται όλε οι διατάξει του κανόνα σύναψη συμβάσεων τη Ένωση. Και εδώ έχουμε θέματα επίση με τι εκταστικέ επιτροπέ σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε πρόσληψη. Και εδώ παρακαλούμε το Ελληνικό συνέδριο να εξετάσει τι βελτιώσει που δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει η αρχή το 2013. Και οι τρει αρχέ έχουν σαφή προκαθορισμένα καθήκοντα. Ωστόσο, αυτό που δεν έχουν. Και αυτό το λέω σε σχέση και με το επόμενο σημείο. Δεν έχουν εντολή στα πλαίσια οδηγιών να επιβάλλουν γραφειοκρατία στα κράτη-μέλη. Η καταξουσιοδότηση πράξης δεν θα πρέπει να επιβάλλουν από μια ελάχιστη προδιαγραμμένη εναρμόνιση μια μέγιστη εναρμόνιση. Και αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον προπολογισμό, αλλά με το μελλοντικό προσωπικό και την πρόσληψη προσωπικού και με την επιθυμία να εκφράζουν άποψη για όλα τα θέματα. Αυτά λοιπόν συνοπτικά είναι σύντομες συγγνωμοδοτήσεις και νομίζω μετά από τις ακροάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού θεωρώ ότι καταφέραμε να συνοψίσουμε τα πιο βασικά σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε αυτές τις παρατηρήσεις πάρα πολύ πάρα πολύ σύντομες και ευσύνοπτες ο τώρα με τους ε, ζήτητες των ε, πολιτικών ομάδων κύριε Φερέιρα ούτε παρίσταται ούτε ότι μπορεί να την καταρχθήσει κάποιος και Ντεμπάκερ Μπάκερ επίσης ε, θέλει τον λόγο δεν ξέρω θέλετε να αντικαταστήσει τον κύριο Όλε Σμιτ μάλιστα. και έχετε τον λόγο Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Όπω ήδη είπαμε, ο, όπως είπατε, μάλλον ο κύριο Ολεσμιτ, ο εισηγητής για την Αλντέα δεν είναι σήμερα εδώ. Είχε στην Σουηδία κάποιε υποχρεώσει, οπότε μιλήσω εγώ για λογαριασμό του. Και θα πρέπει να σα ευχαριστήσω, κύριε Λάγκεν, για αυτά τα οποία συσυντάξατε όσο ως, ε, ως εκθέσεις για την απαλλαγή, συμφωνούμε όσο είπατε και όλη η ομάδα ε, θέλει να δημιουργηθούν ε, αυτές οι τρεις υπηρεσίες και έτσι να έχουμε πιο σταθερές ε, χρηματοοικονομικές αγορέ πιο ασφαλεί, οπότε χρειάζονται και καλύτερο συντονισμό της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αρκετού πόρου, ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία αναθέτουμε και θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα συνομοθέτηση. και επίση είπαμε ότι προσβληματιζόμαστε ότι το Συμβούλιο τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει θελήσει σε αυτέ τι τρει ε, υπηρεσίε να δώσει του πόρου που χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να κάνουν ε, το, το, δουλειά του. Εάν ε, αναθέτουμε επιπλέον αρμοδιότητε σε αυτέ τι υπηρεσίε, όπω κάναμε με μια σειρά οδηγιών και κανονισμών, ε, όπω κάνει το short selling και για τι ε, πιστοληπτικέ αξιολόγηση του, φορεί, πρέπει να του δώσουμε και τι αντίστοιχε, του αντίστοιχου πόρου. Επίση, χρειάζονται προσωπικό στην ε, ΕΣΜΑ και στην ΙΑΤΕ έγινε ε, συρρήκνωση του προσωπικού ακριβώς αντίθετα με ό,τι προβλέπονταν στην αρχή και αυτό έγινε κατά τις διαπραγματεύσεις ε, του προπολογισμού για τη χρήση του 2013. Ήδη οι επικεφαλής των υπηρεσιών έχουν, έχουν επιφυλαχθεί όσον αφορά το, τώρα πώς έχουν, έχουν πρόβλημα, έχουν πρόβλημα να μεταφέρουν και κάποιο είδους πλεονάσματα από τη μία από τη μία ε, ε, χρονιά στην άλλη και επίσης έχουμε και πάρα πολύ ε, προβλήματα όσον αφορά ε, την εμπλοκή και σημεία απόφραξης. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει το Ευρωπαϊκό να κάνει έναν θεώρηση και πώς θα μπορέσει να κάνει την απαλλαγή σε σχέση με αυτές τις ε, υπηρεσίες, θα πρέπει να δούμε καλύτερα τα υπέρ και τα κατά της χρηματοδότησης, αλλά επίσης ε, κάθε επιλογή όσον αφορά τις ε, δυνατότητες της χρηματοδότησης θα πρέπει να τις διευνήσουμε και θα πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο. Τέλος, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πιστεύω θα διαμορφώσουμε μια ευρεία συνένεση και έτσι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε την οποία των προπολογισμών και επίσης το ίδιο να ισχύσει και σαν συνεργασία με τον εισηγητή και τους και εισηγητάς. Κύριε Ντεμπάκη, σας ευχαριστούμε λίγο πρώτα. νομίζω ότι θέλει, θέλει να μιλήσει για τον κύριο Σφέν, τον Σφέν Κιγκόλ. Λάμπερτ, σε συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Όχι, δεν λέω ότι δυσκολεύομαι να σας συγχαρώ, απλώς ε, μου φαίνεται λίγο περίεργο να σας συγχαρώ για τόσο τόσο άρτια ε, ε, έκθεση, γιατί αυτέ οι τρει υπηρεσίε με αυτά τα οποία λέτε σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να του δώσουμε δυνατότητα να συνεχίσουν το έργο του και επίση θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχαμε ένα σωρό διαφωνίε που λέγαμε ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά του, ότι θα πρέπει να γίνουν τα stress test και αυτά αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι ε, αυτές οι υπηρεσίες ουδέποτε είχαν πρικοδοτηθεί ε, με τους πόρους που χρειάζονται για να εκτελέσουν την αποστολή τους. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει και αυτό να τονιστεί. Και κατά τη γνώμη μας, ε, ένας βασικός παράγων ε, αιτία υπηρεσία είναι ο, ο Να μην εξαρτώμεθα δηλαδή όσον αφορά την καλή θέληση των κρατών μελών. Πρόκειται για ομοσπονδιακά θεσμικά όργανα που θα πρέπει και ομοσπονδιακά τέλο πάντων ενωσιακά να, να, να, να πρικοδοτούνται. Μπράβο, Βερνέρ. Οπότε πάντα τέτοια. Ο πρόεδρος. Φιλίπ, ευχαριστούμε. Ο κύριος Κλούτη δεν είναι εδώ. Ούτε κάποιος για να τον αντικαταστήσει. Καλό. Τότε ο Χάνης Πέτερ Μάλιν ας λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις γνωμοδοτήσεις, για την ενδιαφέρουσα δουλειά του. Μία παρατηρήση επιτρέψτε μου σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο συνάδελφος Λάγκε. Όλα αυτά που μας είπατε είναι πάρα πολύ λογικά και κατανοητά διαβάζοντας τις γνωμοδοτήσεις σας. και τις αιτιολογήσεις που ακούσαμε. Όμως κάποια πράγματα μου ακούγονται αρκετά αφηρημένα. Στην βασική ε, έκθεση αναφέρονται συγκεκριμένα τα συγκεκριμένα προβλήματα. Και γι' αυτό εσείς δεν χρειάστηκε να τα αναφέρετε στην γνωμοδότηση. Ή μήπως δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μας, όπως ε, αναφέρεται και στις γνωμοδοτήσεις. Δεν βλέπω κανέναν άλλο το λόγο, να θέλει το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή να απαντήσει. Σας ευχαριστώ να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση και να την απαντήσω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να μην αναφέρονται τα συγκεκριμένα ε, στοιχεία και τα συγκεκριμένα προβλήματα πέρα από την ε, προορισμό της έκτασης της γνωμοδότησης. και στα πλαίσια των περιορισμών ε, που έχει θέσει το Κοινοβούλιο για τις χρηματοδοτήσεις δεν επιτρέπεται να... δεν μπορούμε, δεν χωράνε συγκεκριμένες αναφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συμπεριληφθούν τροπολογίες των συναδέλφων με συγκεκριμένα ε, με συγκεκριμένες αναφοράς, αλλά και εγώ ίδιο ε, χρειάστηκε να κόψω πράγματα γιατί δεν χωρούσαν πολύ απλά στην έκταση του κειμένου. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να μπουν περισσότερα στοιχεία. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Και γι' αυτό και στις τρεις ε, γνωμοδοτήσεις καλό το ελεγκτικό συνέδριο να τα ελέγξει όλα αυτά στις επόμενες εκθέσεις λεπτομερώς. Επιπλέον, από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ε, Αρχή Τράπεζων, Έχουμε μια επιστολή του κυρίου Ρος προς τον κύριο Μάρτιν Σούλτς, όπου μιλάμε για τα θέματα προσωπικού, short selling κτλ. Και αναφέρεται ότι χρειάζεται πιο πολύ προσωπικό. Και νομίζω ότι συνολικά θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ το θέμα αυτό της χρηματοδότησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένος ε, κανόνας, συγκεκριμένη διάταξη. Ήταν μια συμφωνία αυτό το 60-40 και φυσικά οι αρχές χρειάστηκε στην φάση σύσταση του να χρησιμοποιήσουν προσωπικό από τα κρατημέλη, αλλά θέλουν φυσικά στο μέλλον να αποσκοπούν σε μια ανεξαρτησία και κοιτώντας ε, το πόσο αμέριμνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μπορεί και ένα κάτω μέλος μόνο να προβάλλει ένσταση, θεωρώ ότι ως Κοινοβούλιο έχουμε καθήκον να φροντίσουμε για την ανεξαρτησία των τριών αυτών αρχών. ακόμα και αν κάποιες ε, απαντήσεις και ακόμα και αν κάποιες ε, αποφάσεις δεν αρέσουν σε κάποιους. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία. Και αυτό ασφαλώς αποτελεί ε, καταρχάς αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και θα πρέπει να εξαγάγει τα σχετικά συμπεράσματα. Δεν είναι δικό μας καθήκον αυτό, ωστόσο μπορούμε να χρηματοδοτούμε. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ε, δυστυχώς σήμερα λόγω καιρικών συνθήκων δεν είναι άνθρωα η προσέλευση, αλλά όποιος θέλει ευχαρίστως να υποβάλει τροπολογίες για να συμπληρώσει το κείμενο. Ε, ευχαριστώ Βέρνερ. Ε, δεν χρειάζεται χαλαρότητα, χρειάζεται επαγρύπνηση. 29 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. Στις 18 Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 20, ΕΚΟΝ 25 Φεβρουαρίου και στην ε, Αρμόδια Επιτροπή στις 19 Μαρτίου και στην Ολομέλεια τον Απρίλιο ή Μάιο του 2013. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το σημείο και πάμε στο επόμενο. Πάλι εδώ πρωταγωνιστή ο Βέρνερ Λάγκεν Πρόκειται για την οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Κύριε Σεγητά, έχετε το λόγο. Um, äh, Εδώ έχουμε μια διαδικασία συναπόφαση ω τμήμα τη ε, νομοθεσία των χρηματοπιστωτικών αγορών θέμα του Μισελ Μπαρνιέ πέρα από τις τραπεζικές υπηρεσίες οποιασδήποτε φύσεως, ε, θα πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου και θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Έγινε μια συζήτηση για το κατά πόσο αυτό είναι σωστό, είναι απαραίτητο, αναγκαίο να οριστεί μια ελάχιστη εναρμόνιση, κατά πόσο να πρέπει να ξεπεραστεί αυτή η ελάχιστη εναρμόνιση μετά από διεξοδικές διαπραγματεύσεις και πολλές πολλές προτάσεις που διατυπώθηκαν, θεωρώ ότι η ελάχιστη εναρμόνιση είναι ο σωστός δρόμος. Γιατί κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις θεωρούν ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν αποτέλεσε και το μελετησέριτος όπως παρουσιάζεται συχνά. Υπάρχει μία εξαίρεση, τα μακροπρόθεσμα προϊόντα ασφάλειας ζωής που φυσικά δεν μπορούν να συγκριθούν με μια ασφάλεια ταξιδίων, ακύρωση ταξιδίου. Αυτό εξαρτάται από την αγορές αλλά και από το κόστος. Θα πρέπει ασφαλώς να ε, προστατεύσουμε πιο πολύ τον καταναλωτή για να αντιμετωπίσει και τις εξελίξεις στις αγορές. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση αυτή θα πρέπει να αξιολογηθεί με διαφορετικό τρόπο. Στην έκθεσή μου, στο σχέδιο έκθεσης, περιλαμβάνω κυρίως τεχνικά ζητήματα. Να, να ευχαριστήσω τον κύριο Φαν Έσ από τη Γραμματεία που με βοήθησε πάρα πολύ. 109 τροπολογίες, εκ των οποίων μια σειρά ε, επιτεχνικών λεπτομεριών, αλλά και κάποιες επί της ουσίας. Το θέμα λοιπόν είναι και κάποιες ασάφειες, οι οποίες θα πρέπει να διευκρινιστούν. Γι' αυτό λοιπόν ε, έχουμε, θέματα, έχουμε τη συζήτηση μπροστά μας, στήφονται θέματα μετάφρασης, στήφονται θέματα υπολογισμού σε βάθος χρόνου. σε ό,τι αφορά τις ε, ασφάλειες πίστοσης ακολουθείται η απλοποιημένη διαδικασία. Θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει ασφαλώς. Αλλά συνολικά πρέπει να πω ότι υπάρχουν επτά βασικοί τομείς. Και με αυτούς μπορούμε να πετύχουμε την ελάχιστη εναρμόνιση. Παιδί εφαρμογή καταρχάς. Εδώ θα πρέπει να ισχύουν ίση όρια ανταγωνισμού αυτό είναι ο σκοπός της Επιτροπής και γι' αυτό προτείνει πώληση ασφάλισης ε, ε, και επέκταση του πεδίου εφαρμογή στην πώληση ασφαλίσεων. Εδώ έχω κάποιες ε, αμφιβολίες και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση περιπτώσεων ζημιών γιατί θα σήμαινε αυτό τεράστια επέκταση και θα έδινε την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αργότερα βάσει ενός ε, κενού, αν θέλετε, αμφισβητούμενου κενού, να προτείνει άλλες διατάξεις. Άρα, εγώ δεν θα θέλω να συμπεριληφθούν αυτά σε ό,τι αφορά τις ταξιδιωτικέ ασφαλίσει και αντασφαλίσεις, σε ό,τι αφορά ενοικίε αυτοκινήτων σε επικουρική δραστηριότητα θα πρέπει να προταθεί μια ρύθμιση εξαίρεσης μακότητας. Κοιτώντα την ταξιδιωτική αντασφάλιση, ο τομέα μα λέει ότι 100, 140 εκατομμύρια το χρόνο αφορούν χαμηλά ποσά όπου το κόστος ενδεχομένως θα αποτελούσε το ίμιση της ασφάλισης, αλλά κάθε καταναλωτής ε, που κλείνει ένα ταξίδι 3.000 ευρώ για παράδειγμα είναι διατεθειμένος ε, να πληρώσει για 30 ευρώ για ασφάλιση χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία. Εδώ είναι το θέμα της αναλογικότητας που τίθεται και γι' αυτό ε, ζητούμε να εξαιρεθεί. Ύστερα, δεύτερο θέμα, εγγραφή και απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής. Ο τομέας, το παιδί εφαρμογή ε, επεκτείνεται σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους. Και γι' αυτό τίθεται το ερώτημα για το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει εκ νέου εγγραφή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του προσωπικού τους. Θεωρώ ότι μια νέα εγγραφή αυτών δεν είναι απαραίτητη. Μία άλλη αλλαγή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως επικουρική δραστηριότητα οι προηγουμένες προϋποθέσεις. Αυτό υποστηρίζεται. Αλλά τύφονται θέματα ε, ευθύνης αν κάνει ένας τρίτος μία σύμβαση σε περίπτωση ε, που υπάρχουν ε, διαφορές, αυτό τίθεται ως προβληματικό. Άρα, μιλάμε λοιπόν για ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείε ενοικίαση αυτοκινήτου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ προβλέπει απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής, αλλά εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η οδηγία δεν θα ισχύει για, τα για τους τρεις αυτού τομείς. Και θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν το άρθρο 4 σε ό,τι αφορά την απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να διευκρινιστεί. Έχουμε επίση τι επαγγελματικέ και οργανωτικές απαιτήσει στο άρθρο 8. Η Επιτροπή πρότεινε συνεχή και διαρκή επαγγελματική κατάρτιση για την εξασφάλιση των κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων των διαμεσολαβητών. Αυτό ασφαλώς ε, το καλωσορίζουμε. Το ερώτημα ωστόσο είναι ποιος θα είναι υπεύθυνο. Ε. Είναι θέμα αυτορύθμισης και αυτοοργάνωσης των κρατών μελών ή όπως στην προηγούμενη έκθεση θέλουμε ένα εκτεταμένο ετήσιο μητρό όπου ο, όλοι οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις εγγραφής τους με κυρώσεις. Είναι αυτό αναπαραίτητο. Εγώ πιστεύω πως όχι, γιατί σε ό,τι αφορά τα ελεγκτικά συστήματα τα οποία ισχύουν στα κρατημέλη, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν και θα πρέπει να τίθενται ε, επαγγελματικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ως προς τις, ε, τα προσόντα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και θέματα αμοιβέ αναγνώριση. Να σα αναφέρω τη Γαλλία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, προδιαγράφεται και είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου μάστερ. Δεν χρειάζεται πρακτική εμπειρία. Σε άλλες χώρες χρειάζεται πρακτική εμπειρία και μάλιστα εξετάσεις. Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα και αυτό θα ήθελα να το συμπληρώσω γιατί δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει κάθε χρόνο τι γίνεται σε ό,τι αφορά την ε, ε, αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ χωρών. Για παράδειγμα, η Allianz και η Άξα ως μεγάλες επιχειρήσεις και εταιρείε ασφάλειας. Προσφέρουν τα προϊόντα ανά χώρα, ανά μέλος. Ουσιαστικά σπάνια υπάρχουν ταυτόσιμα προϊόντα τα οποία αναπαρέχονται σε όλες τις χώρες, άρα υπάρχει ο κίνδυνος εδώ για το Γάλλο καταναλωτή, αν του προσφέρει ένας, ε, μια γερμανική εταιρεία ένα προϊόν, να μην ισχύουν οι, δύο, οι ίδιοι όροι. Το ίδιο ισχύει και αντιστροφά ασφαλώς. Και εδώ τι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε περίπτωση σύγκρουσης, αυτό αποτελεί και η βασική φιλοσοφία της ενιαίας αγοράς, σε περίπτωση αμφισβήτησης και ε, σύγκρουσης να υπάρχουν ίδιοι όροι με μια μεταπαιδική φάση. Ύστερα έχουμε τα κέντρα επαγγελματική κατάρτισης. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο σε ό,τι αφορά την εθνική πιστοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισής τους. Γιατί δεν είναι πιο δύσκολη η πιστοποίηση κάθε ενός διαμεσολαβητή. Είναι πάρα πολύ, πάνω από ένα εκατομμύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό θα συνεπαγόταν τεράστιο γραφειοκρατικό άχθος, το οποίο ούτε είναι αναγκαίο, ούτε είναι αναλογικό. Ύστερα, έχουμε συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια. Εδώ έχουμε πολλές τροπολογίες για το άρθρο 17. Η Επιτροπή προβλέπει υποχρέωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών να χρησιμοποιούν τη βάση για το ακριβέ ύψο τη αμοιβή του, καθώ και το ακριβέ ύψο τη μεταβλητή αμοιβή των υπαλλήλων πολίσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα ασφάλεια ζωή προβλέπεται η άμεση εφαρμογή τη υποχρέωση αυτή με την έναρξη ισχύω τη οδηγία, ενώ για την πώληση προϊόντων ασφάλισης εκτό ασφαλιών ζωή προβλέπεται αρχικά να ισχύει κατόπιν ετήματο με μεταβατική περίοδο 5 ετών. Αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και ξέρω ότι είναι πολύ διαφορετικέ οι απόψει που επικρατούν στο Κοινοβούλιο σχετικά και της δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή μάλλον μεταβίβαση σε... της αμοιβής αυτής. Και σε ό,τι αφορά θέματα γνωστοποίησης. Το θέμα όμως είναι Τι προμήθεια θα ε, παίρνει ο διαμεσολαβητής ή η ποιότητα του προϊόντος. Δεν μπορεί το θέμα μας να είναι αν πήρε 200 300 ευρώ ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Αυτό θα οδηγήσει ουσιαστικά, σε, θα οδηγούσε σε ανταγωνισμό μεταξύ των διαμεσολαβητών και όχι σε βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Το θέμα είναι επίση και αυτό δεν αναφέρεται, να βρούμε μια, ένα συμβιβασμό για τι μακροπρόθεσμες ασφάλειες ζωής. Να αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία ή ποσοστά του συνολικού όγκου. Αυτά είναι τα πιο βιώσιμα, αν θέλετε, προϊόντα, τα οποία προκαλούν και τα πιο υψηλά, τις πιο υψηλές δαπάνες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει εντατικά. Θα πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν έχω κάνει σχετικές ε, προτάσεις, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει μια γραμμή συμβιβασμού. Έχουμε επίσης διασταυρούμενες πωλήσει. Άρθρο 21. η Επιτροπή προβλέπει ότι οι ασφαλιστικέ υπηρεσίε και τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρονται ω δέσμοι θα πρέπει να μπορούν να προσφέρονται και χωριστά. Αυτό υπερβαίνει την αντίστοιχη ρυθμίση τη οδηγία MIFID 2 και θα μπορούσε να έχει ω αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να προσφέρονται οικονομικέ για τον καταναλωτή δέσμε προϊόντων. Για το λόγο αυτό, το άρθρο 21 θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε οι καταναλωτέ να ενημερώνονται μόνο σχετικά με το αν είναι δυνατή η αγορά χωριστών στοιχείων δέσμη. Η συνάδελφο Στήλερ στην ΙΜΚΟ πρότεινε κάτι διαφορετικό υπερβαίνει και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, εκφράζει γενικά αμφιβολίες για τις διασταυρούμενες αυτές ασφάλειες. Εδώ, κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Περιμένω να λάβω και τις τροπολογίες των συναδέλφων. για να μην υπάρξει και επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος. Αν κάποιος παίρνει ένα δάνειο και ασφάλεια πίστοσης, μαζί με το δάνειο, αυτό θα ήταν πρόβλημα, γιατί θα ε, υπαγόταν αυτό στις ε, πωλήσει προϊόντων, γιατί είναι προϊόν η πίστοση και αυτό θα επιβάρυνε τον καταναλωτή. Σκοπός είναι να λαμβάνει την πληροφόρηση ο καταναλωτής ότι μπορεί να αγοράσει και ξεχωριστά κάποια ασφαλιστικά προϊόντα. Ύστερα, τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. Η Επιτροπή εξετάζει πρόσθετε απαιτήσει προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα λεγόμενα PRIPS. Η κυρία Μπερές θέλει αυτά να τα ρυθμίσει με εξατομικευμένο τρόπο. Δεν θέλει να υπάρχουν γενικά πακέτα, αλλά και κάθε προϊόν να να υποβάλλεται ξεχωριστό πακέτο. Θεωρώ ότι αυτό θα προ... προκαλέσει υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση και για τους ε, ασφαλιστές και για τους ε, καταναλωτές. Σημαντικό είναι να ρυθμιστούν τα θέματα ευθύνης. Να υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές σε ό,τι αφορά την ευθύνη. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Να μην υπάρχουν απαγορεύσει. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται δηλαδή οι διατάξεις. Αν κάποιος για παράδειγμα έχει λάστιχα τα οποία δεν θεωρούνται καλά σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο και προκαλέσει ατύχημα σε γερμανικούς δρόμους έμεσα να φροντίζει η ασφάλειά του, να μην τον ασφαλίζει. Να μην είναι δηλαδή εξατομικευμένη περιγραφή, να υπάρχει μάλλον περιγραφή των προϊόντων. Γιατί ιδάλλως θα έπρεπε να ελέγχουμε κάθε μια μεσολαβητή ξεχωριστά. Και αυτό δεν θα οδηγούσε στην ε, μείωση της ε, γραφειοκρατίας. Τώρα, η απαγόρευση που προτείνεται για τις προμήθειες. Αυτό υπήρξε σε κάποια κρατημέλη. Δεν αξιολογήθηκε θετικά μέσα από έρευνες. Μάλλον ως αρνητικό αξιολογήθηκε σε ό,τι αφορά την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων στον πληθυσμό. Και το λοιπόν ε, αμφιβάλλω κατά πόσον θα βελτιώσουν την προστασία του καταναλωτή. Έχουμε το θέμα των προσόντων τώρα. Το ανέφερα. Εδώ χρειάζεται αμοιβαία αναγνώριση. Και αυτό αφορά και την περαιτέρω κατάρτιση. Δεν χρειάζεται όμως ε, η ε, ίδιες προδιαγραφές για όλους. Τελευταίο σημείο από πλευρά μου, οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Η Επιτροπή προβλέπει σειρά κατά εξουσιοδότηση πράξεων σε τομείς οι οποίοι αφορούν σημαντικά θέματα της οδηγία, ορισμό των κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων των διαμεσολαβητών, κριτήρια για τη βάση πολιτισμού τη προμήθεια, μέτρα για την αποτροπή, τη ρύθμιση και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων συμφερόντων, υποχρεώσει, ενημέρωση και εν των πελατών, εγώ θεωρώ ότι γενικά το θέμα αυτό είναι αμφισβητούμενο, γιατί δεν εξυπηρετεί το στόχο που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλουμε να πετύχουμε, που είναι η ελάχιστη εναρμόνιση. Όχι, εξυπηρετούν το σκοπό από το παράθυρο που προσπαθεί να μπει, της μέγιστης ε, εναρμόνισης. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να διαγραφεί αυτό το ζήτημα και να αποφασίζονται αυτά μέσω διαδικασίας συναπόφασης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Να σας υπενθυμίσω ότι οι πέντε πρώτες ε, οδηγίες που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέχουν αντιφάσεις με το πρωτογενές δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θέλω να περιοριστούν αυτά στο ελάχιστο. Γιατί το θέμα δεν είναι η γραφειοκρατική επιβάρυνση. Όχι, το θέμα είναι να καταλήξουμε σε, ένα καλό, σε μια καλή ρυθμίση. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Ο γραφειοκρατικός έλεγχος ό,τι αφορά τις ενστάσεις και τις καταγγελίες αναφέρεται, όπως μου είπαν, στο ΑΙΟΠΑ ότι όλες οι καταγγελίες θα πρέπει να συλλέγονται και όλες οι καταγγελίες θα πρέπει να αξιολογούνται, να καταγράφονται και να απαντώνται με γραφειοκρατικό τρόπο από τις 18.000 καταγγελίες που ε, προέκυψαν πέρσι. Αυτά τα στοιχεία αφορούν τη Γερμανία. 18.000 καταγγελίες στη Γερμανία προς την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή. Μόνο 6, μόνο 6 από τις 18.000 αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Όλες οι υπόλοιπες έχουν να κάνουν το περιεχόμενο των ε, ασφαλιστικών προϊόντων που δεν αποτελούν θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της ε, οδηγίας αυτής. Μιλάμε για 6 στις 18.000 καταγγελίες. Άρα, για να αποφύγουμε το γραφειοκρατικό αυτό άχθος, νομίζω ότι δικαιολογούνται οι κατεξουσιοδότηση πράξεις. Γι' αυτό λοιπόν συνάδελφοι σας παρακαλώ ελάχιστη εναρμόνιση όσο το δυνατόν λιγότερες πράξεις κατεξουσιοδότηση και να τηρούνται και να γίνονται σεβαστά τα διαφορετικά εθνικά συστήματα σε ό,τι αφορά την περαιτέρω εξέλιξη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για τις πολύ αναλυτικές ε, τεχνικές ε, επεξηγήσεις. Ο κύριος Σάντσος Πρεσέδο είναι στην Επιτροπή Αλίας. Ε, δεν είναι εδώ λοιπόν. Θα, θα, δώσω τον, θα δώσω τον λόγο στον νέο εκπρόσωπο του κύριου Όλε Σμιτ. Ο Όλε Σμιτ είναι σήμερα στη Σουηδία και δεν μπορεί να παραστεί σε αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό θα μιλήσω εξ ονόματός του. Ευχαριστώ τον κύριο Λάγκεν για την έκθεσή του. Ο κύριος Όβιος Σμιτ θέλει να κάνει κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Η πρόταση της Κομισιόν είναι σημαντική πρωτοβουλία για αυξανόμενο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και για την ολοκλήρωση της αγοράς μέσα στην ενιαία αγορά. Χρειαζόμαστε ανοιχτή, ανοιχτές χρηματαγορές και υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών για να ξανακερδιθεί η εμπιστοσύνη τους. Επειδή είναι κατακαιρματισμένη η αγορά στα διάφορα κράτη-μέλη, μια ελάχιστη προσέ... η προσέγγιση ελάχιστη εναρμόνισης είναι κατάλληλη. Το επίπεδο όμως προστασίας των, των επενδυτών θα πρέπει να αυξηθεί για να μειώσουμε την ανάγκη για διαφορετικά εθνικά μέτρα. Όπως υπόθηκε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ο ΣΜΙΤ πιστεύει ότι είναι σημαντικό να κρυφθεί υπόψη η φύση των συμβάσεων αυτών, ασφαλιστικών συμβάσεων, σε σχέση και σε αντιδιαστολή με τα επενδυτικά προγράμματα. Εδώ έχουμε και τα, τις ασφαλίσεις σε επενδυτικά προϊόντα. Θα πρέπει να βασιστούμε πάνω στην IMD, δηλαδή στην οδηγία για τις ασφαλιστικές συμβάσεις και όχι στη MIFID. Ο κύριος Λάγκεν τονίζει διάφορα βασικά θέματα και μιλάει για σημαντικές αλλαγές που είναι ευπρόσδεκτες. Ε, με βάση την άποψη του Όλε Σμιτ, όμως πρέπει να ενισχύσουμε την προστασία των καταναλωτών. Η ποιότητα των συμβουλών είναι σημαντική. Ε, στο παρελθόν υπήρχε προβλήμα, υπήρξαν προβλήματα με τις πωλήσει στη Σουηδία και σε όλη την Ευρώπη. Και θα πρέπει να καλύπτουμε πάντα τις ανάγκες των επενδυτών. Οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν προϊόντα με βάση σωστές συμβουλές. Το άρθρο 17, στο άρθρο 17 οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πάντα τη σύγκρουση συμφερόντων όταν για την αμοιβή, για τις αμοιβές. Πρέπει να υπάρχει πολιτική διαφάνεια των αμοιβών για να ε, έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές στον ενδιάμεσο, θα πρέπει να γνωρίζουν όλα τα χρηματικά κίνητρα. Ακόμη και αν ο καταναλωτής δεν ζητήσει αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να του παρέχονται θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνε από πλευρά τη Κομισιόν που να προστατεύουν όλου του καταναλωτέ στην Ευρώπη. Ε, Πλήρη διαφάνεια, αποκάλυψη των πληροφοριών, αυτά είναι απαραίτητα. Ο ενδιάμεσο θα αποφασίσει αν θα χρησιμοποιεί όχι τον όρο ανεξάρτητο. Οποιοδήποτε ενδιάμεσο θέλει να πληρώνεται μέσω ε, προμηθειών μπορεί να επιλέγει όχι τον όρο ε, ανεξάρτητο ή όχι. Η Κομισιόν λοιπόν θα μπορεί να επιλέγει ε, τι είδου συγκρούσει συμφερόντων υπάρχουν. Ε, επίσης η διαχείριση των απαιτήσεων. Συμφωνούμε να, με τον κύριο Λάγκεν να αποκλείσουμε τις απαιτήσει και να διαγράψουμε, το διαγράψουμε αυτό από το άρθρο 4 για να υπάρχει η ισοτιμία. Ε, πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τους υπόλοιπους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές. Ο Φιλίπ Λαμπέρ. Σε ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι αντικαθιστά τον Σβέν έχει το Ευχαριστώ πρόεδρε να αρχίσω ευχαριστώντας όλους τους αδελούς που είναι εδώ. θα μπορούσα να και περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι είσαστε, εγώ κάνω το πόλο το ΕΦ, οπότε ελπίζω ότι θα μπορέσω να αρχίσω την προσοχή σας μέχρι ότου τελειώσει η συνεδρίαση. Οπότε, να μην θεωρείτε ότι χάσατε το χρόνο σας σήμερα το απόγευμα. Πέραν αυτών, Για άλλη μια φορά συμβαίνει και ανησυχώ ότι σύμφωνα με τον Βέρνερ Λάγκεν. Ναι, θέλουμε τέτοια την ελαχίστη δυνατή εναρμόνιση, τέτοια προσέγγιση και θα πρέπει να έχουν πιο ψηλά τον πύχη επομένω τα κράτη-μέλη και όπω και για άλλα θέματα θέλουμε αυτό ο ελεύθερο κοινό προγραμματή όμω να είναι ψηλούτσικο. Άρα θα πρέπει να, να, να έχουμε υψηλέ προσδοκίε γιατί τελικά αυτό το οποίο εδώ πέρα αποτελεί το κίνητρο είναι η προστασία του καταναλωτού. Οπότε γι' αυτό και έχουμε και κάποιες σχετικές τροπολογίες. Μάλιστα, όντως, είναι ορθή κίνηση η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα δίκτυα του καταναλωτή. Αλλά νομίζω θα μπορούσαν να γίνουν και ακόμα περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση σε αυτή την έκθεση. Και όσον αφορά τώρα την ασυμμετρία της πληροφορίας, ε, συμφωνώ με τα περισσότερα που ανέφερε ο Φιλίπ Ντεμπάκερ όσον αφορά την διαφάνεια, τα συστήματα της αντιστάθμισης και έτσι να δούμε πώς θα μπορούμε να τονώσουμε τον ανταγωνισμό και πώς θα έχουμε ποιοτικέ συμβουλές. Οπότε, πώς θα γίνει. Θα μπορούσε κάτι να γίνει. Έχουν αυτοί οι μεσίδες συνδιάμεση τις δεξιότητες, τα προσθέτω που χρειάζεται και επομένως έτσι να έχουν ψηλότερο επίπεδο. Κάτι άλλο επίση για το οποίο θα κατεβάσουμε τροπολογία είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή ή των Ευρωπαϊκών Ευρωπαϊκών Αρχών και τέλο δε θα πρέπει να δούμε πώ θα είμαστε όσο γίνεται πιο συνεπεί όσον αφορά αυτού του είδου του κανονισμού ε, και άλλου όπω το MIFID. Θέλουμε να είναι αποτελεσματική η νομοθεσία. Δεν θέλουμε να υπάρχει πολυνομία και ε, γραφειοκρατία Γι' αυτό και προς τα εκεί θα κρατείνουν οι τροπολογίες μας. Αυτά για το παρόν νομοθέτημα. Ο πρόεδρος, Φίλιπ, σε ευχαριστούμε. Άσλι Φόξ. Όχι, δεν είναι εδώ. Κάποιος για συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Ούτε ο κύριος Πρασέα Πρασέδο έχει έρθει. Άρα, έτερος, ουδής, Σιμών. Κύριος Σάιμον. Äh, αυτό που θέλω να πω αφορά τα όσα ακούσαμε τον κύριο Ντεμπάκερ. Δεν ξέρω, αυτό, αν εγώ δεν κατάλαβα καλά. Δεν κατάλαβα καλά τι βέβαια, ποια είναι η γνώμη του. Όσον αφορά αυτούς τους ανεξάρτητους συμβούλους. Αυτούς που ε, αυτό που μπορούν κάποιοι μεσίτε να, να, να αυτοαποκαλούνται. Και αυτό να ισχύει ανεξαρτήτω του αν έχουν κάποιο προμήθεια. Γιατί εγώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε εισπράττει κάποια προμήθεια, ε, τότε πάβει να είναι ανεξάρτητο. Μα αν παίρνετε προμήθεια, ζείτε από αυτήν, άρα εξαρτάστε από αυτήν. Αν κάποιο θέλει συμβουλέ και θέλει εξάρτητε πληροφορίε, θέλει πραγματικά κάποιο τέτοιο πρόσωπο. Αν όμως θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα που να βασίζεται σε, σε, σε προμήθεια, θέλουμε να διατηρηθεί ένα τέτοιο σύστημα, τότε αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι οι συμβουλές τις οποίες δέχεται δεν είναι δωρεάν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Πρόεδρος. Έχω αυτή την παρατήρηση. Πρώτη κάτι το οποίο το συζητήσαμε στον Ρωτονίφιλ. Και είχαμε καταλήξει και σε ένα συμβαστικό κείμενο για την Ολομέλεια. Δεν θέλω να πει λεπτομέρειε, αλλά στα γερμανικά έχετε δύο λέξει σχετικά και εμεί μόνο μία στα γαλλικά. Έχω δύο τέλο πάντων λέξει που αποδίδουν την λέξη ανεξάρτητο, αμερόληπτο τέλο πάντων. Οπότε αυτοί οι μεσίδε θα πρέπει να αποδείξουν ότι όντω είναι ελευθέρωτο το επαγγελμά του, ότι είναι ανεξάρτητοι, ότι δεν, δεν, δουλεύουν στο πλαίσια ενό ομίλου. Να το πρόβλημα αυτό, όπω το, το, αναφέρατε. Και γι' αυτό και στην Μιφίντ και στο κείμενο της Ολομέλειας είχαμε πει ότι ε, η Συμβουλή όχι ανεξάρτητη, αλλά κάποιο σύμβουλο ο οποίο είτε επί τη βάση προσωπικών γνώσεων ε, δίνει αυτά επί τη βάση των όσων ξέρει, οπότε και έτσι αμείβεται αντιστοίχω και κατόπιν ο σύμβουλος ισχυρίζεται ότι ό,τι είπε το είπε ανεξαρτήτως από τις επαφές, τις γνώσεις του με αυτόν από τον οποίο προέρχεται το χρηματιστηριακό προϊόν. Και γι' αυτό σε εκείνη την περίπτωση είχαμε πει ότι δεν δικαιούται κάποια αμοιβή για τη MIFID. Και στο και είδαμε ότι υπάρχει εκεί ένα σφάλμα στη, στο κείμενο εκείνο και στον τρίλογο το είχαμε διορθώσει. Είπαμε ότι εκείνο ο οποίο υπάρχει ανεξάρτητε συμβουλέ δεν μπορεί να αμοιβεται καθόλου. Ούτε καν από το σύμβουλο του, το οποίο βέβαια δεν στέγει. Αυτό διορθώθηκε τελικά στον τριμερή διάλογο. Φυσικά και μπορεί να ανέβεται από τον πελάτη του. Αυτό ισχύει στη Γαλλία. Έχουμε κάποιον μεσίτη με 3.000 πελάτες και ένας του, του, πληρώνει δυναμιδή και μόνο ένας από αυτού του αναδρομικό σύστημα. Κύριε Σκίνερ, ναι, σας ευχαριστώ. Αυτό το περάτε για αμοιβή ή για μεσητεία, προμήθεια, πολύ σημαντική. Κυρίως γιατί έχουμε δεκάδες χιλιάδων που προσπαθούν έτσι να, να ζήσουν από τους πελάτες τους. Θα πρέπει επομένω να βρούμε μια λύση που να λαμβάνει όλες τις πλευρέ υπόψη. Τελικά, στο μέλλον θα πρέπει να εξετάσουμε κανείς από πού αγοράζει ασφαλιστήρια. Πολλές φορές βγαίνουν στο ίντερνετ, συγκρίνουν τις τιμές. Και θα πρέπει μετά ο καθένας μόνος του να βρει ποια λύση πιο ασφαλιστήριο πλεονεκτή. Τελικά αυτοί οι μεσίτες των πάντων είναι μια χαρά επαγγελματίε, αλλά ζουν από αυτές τις αμοιβέ ή τις προμήθειες. Δεν διάβασα όλες τις λεπτομέρειες, αλλά όμως είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει για να έχει καλή οργάνωση η ασφαλιστική αγορά να βρουν τους σωστή και στην Αμερική όπως ξέρετε οι αντίστοιχοι μεσίτες εξαρτώνται από αυτούς που έχουν συμφέρον. Συμφέρονται τόσο συγκεκριμένα στην ασφαλιστική αγορά. Θέλω να πω ότι ό,τι λύση και να δοθεί θα πρέπει να λάβει επόμενο υπόψη ο αυτοριστικής αγορά. Ο κύριος Σάντσος Πρεσέδο έρχεται με βήματα χήμου, λένε. Έχουμε όλα τα συστήματα για να εντοπίζουμε τους βουλευτές. Έχουμε GPS και ξέρουμε πολύ καλά ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο καθένας. Ας περιμένουμε τον κύριο Σάντσο Περσέδο. Ε, η κυρία Μπερές έρχεται για την επόμενη έκθεση. Δεν θα κάνουμε κανένα διάλειμμα. Ε, όταν τελειώσουν το λόγο οι ευρωβουλευτές, πάρουν όλοι το λόγο, θα δώσω το λόγο στον Βέρνερ. Τέλο πάντων, Βέρνερ, μπορεί τώρα να μιλήσεις και μετά θα δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο, τον Σάντζες Περσέντο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Τα αμφισβητούμενα θέματα τα αναφέρατε όλοι να ευχαριστήσω τον Πίτερ Σκίνερ που αναφέρθηκε στο θέμα του διαδικτύου και τα προβλήματα με το ίντερνετ. Ο, η κυρία Στίγλερ στην ΕΜΚΟ ε, πρότεινε να προδιαγραφούν υποχρεωτικές συγκρίσεις τιμών. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο, αλλά εγώ τι πιστεύω και ότι φαίνεται ότι προσεγγίζουν τιμές στο διαδίκτυο αλλά πρώτα υπάρχει μια διαβούλευση και μετά γίνεται η αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος. Και έρχεται και ο συνάδελφος. Σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις για τις αμοιβέ. Σημαντικός τομέας αυτός κάποιοι τομείς όπως ε, η βιομηχανικός τομέα για παράδειγμα, η ναυσίπλο ή ναυπηγικές εταιρείε δραστηριοποιούνται έντονα εδώ. Και δεν ε, μπορούμε να προκαλέσουμε κατακαιρματισμό σε ό,τι αφορά τις αμοιβέ. Δεν θα ωφελήσουμε και τον καταναλωτή. Να πω επίσης ότι οι εκθέσεις διατίθενται σε όλες τις γλώσσες. 6 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για κατάσταση τροπολογιών. Ο κύριος ε, Βίξτρομ ζήτωσε να παραταθεί αυτή η ημερομηνία. Θα μπορούσαν να αποταθούν ένα-δυο μέρες. 7-8 Φεβρουαρίου το αργότερο ωστόσο. Και το θέμα του πώς θα συμπεριληφθεί η ΙΜΚΟ δεν έχει ακόμα αποφασιστεί αυτό, από το Συμβούλιο ξέρω ότι το θέμα αυτό της διαμεσολάβησης ε, ασφαλιστικών προϊόντων έχει τεθεί σε τεχνικό επίπεδο, αλλά δεν αποτελεί προτεραιότητα της Ιρλανδικής Προεδρίας ως τώρα. Όσο πιο γρήγορα ολοκληρώσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις μας, τόσο πιο άμεσα μπορούμε να αναγκάσουμε το Συμβούλιο να δράσει ακόμα και άμα δεν το επιθυμεί. Αυτά λοιπόν πριν πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι. Κύριε Αντολίνο, ε, σας παρακολουθήσαμε απευθείας ε, στις ε, οδηπορίες σας ε, μέσα στο Κοινοβούλιο. Έχετε κατεξαίρεση το λόγο τώρα μετά τον εισηγητή. Ναι, στην Επιτροπή Αλίας ήμουν. Και εκεί είχαμε την πολύ σημαντική συμφωνία με τη Βρετανία και ήμουν εγώ εισηγητής. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκεν. Δεν θέλω να πω τίποτα σαν αντίρρηση, απλώς να πούμε κάτι για τις τροπολογίες, είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτές τις εκθέσεις. Οι τροπολογίες του κυρίου Λάγκη είναι πολύ σημαντικές. Αυτό το μητρό, το πρωτόκολλο, την επαγγελματικότητα πρέπει να διακρίνει αυτά τα πρόσωπα. Τι θα κάνουμε για τη σύγκρουση συμφερόντων. Και εν πάση περιπτώσει, ο ρόλος αυτών των επαγγελματιών έχει να κάνει πολύ με το μάρκετινγκ. Ξέρω ότι κουράστηκε πολύ ο συγητής. Γι' αυτό και εγώ στις τροπολογίες μου θα διαπνέομαι από όσο γίνεται περισσότερο πνεύμα συνεργασίας και έτσι να διεκπαιριώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα το θέμα. Βέβαια, θες να απαντήσεις αυτούς όλους επένους. Να σας ευχαριστήσω και εγώ να σας πω ότι θα συνεργαστούμε όσο το πνευμόν και όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κανένας άλλος να πάρει το λόγο. Να σας διευκρινίσω ότι η Επιτροπή ΙΜΚΟ ζήτησε να χρησιμοποιήσει το άρθρο 50 για την ενισχυμένη συνεργασία. Μελετάτε το θέμα και ο πρόεδρος της Επιτροπής θα δώσει τη γνωμοδότησή του 31 Ιανουαρίου ή 7 Φεβρουαρίου. οι ημερομηνίε. Καταθέτουμε τι τροπολογίε 6 Φεβρουαρίου στι 12 το μεσημέρι. Θα τι εξετάσουμε 25-26 Φεβρουαρίου του 2013. Θα, θα ψηφίσουμε στις 26 Μαρτίου του ΕΚΟΝ και στην Ολομέλεια του Μαΐου του 2013 θα εξεταστεί το θέμα. Ο κύριος Πρεσέδο ζήτησε μια μικρή ε, αναβολή για τις ε, τροπολογίες. Επιμένετε κύριε Σάντος Πρεσέδο. Βέρνερ. Δεν το έλεγξα. Δεν έχει αναβληθεί η συνάντηση πριν από το Πάσχα, 27 Μαρτίου. Δεν έχει αναβληθεί, δεν έχει αλλάξει αυτή η ημερομηνία. Μήπως το θυμάμαι λάθος. Okay, good. später. Μάλιστα, καλά. Το κοιτάμε πιο αργά. Ποιο έχει ποιο μετά την φάση κάποια άλλη στιγμή. Ωραία, σταματάμε λοιπόν εδώ για αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο. Είναι εδώ η συγγήτρια. Και βλέπουμε ένα μεγάλο πλήθος ε, που θέλει να παρακολουθήσει αυτό το σημείο. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο που αφορά τις ε, ουσιαστικές πληροφορίες και τα έγγραφα με βασικές πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα. Κύριε Μπερές, έχετε το λόγο. Επιτέλους, δίνω εγώ ως πρόεδρος το λόγο στην πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Σας εκδικούμε κυρία Μπέρες. Σας συγχαίρω για την προαγωγή σας ως πρόεδρος στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Χαίρομαι που θα, θα παρα... παρουσιάσω αυτό το σημείο. Α, είπα προηγουμένω, ή μάλλον ξέχασα να πω προηγουμένως ότι μόνο χάρη στην ηλικία μου πήρα αυτή η θέση. Θέλω να σας παρουσιάσω μετά από μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έγινε στα τέλη του 12 σήμερα αυτό το σχέδιο έκθεσης για την πρόταση της Κομισιόν για τα επενδυτικά προϊόντα για τα δεσμοποιημένα επενδυτικά προϊόντα. Πρόκειται για το αγγλικό ακρονίμιο PRIPS, Package Retail Investment Products, δεσμοποιημένα επενδυτικά προϊόντα που προορίζονται για το λιανεμπόριο. Θέλω και το δικό μου κείμενο και το κείμενο του Βέρνερ να προχωρήσουν παράλληλα, γιατί δεν πρέπει να γράψω άλλο εγώ και άλλο Βέρνερ στα δύο κείμενα, γιατί και τα δύο μιλούν για την προστασία των καταναλωτών. Στο σχέδιο έκθεσης που σας έχω ήδη παρουσιάσει, σας προτείνω ένα σημαντικό αριθμό τροπολογιών. Μιλάω για 64 τροπολογίες. Θα σας παρουσιάσω την γενική φιλοσοφία τους. Η πρόταση της Κομισιόν έχει σαν σκοπό να ενημερώνονται οι αποταμιευτές και εκείνοι που αγοράζουν τέτοιου τύπου ε, δεσμοποιημένα επενδυτικά προϊόντα, packaged, πρόκειται για μια αρχή η οποία διαπνέεται από την ιδέα της προστασίας των καταναλωτών. προκειμένου να αποκαταστήσουμε και με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους στην αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Στις τροπολογίες σας προτείνω ε, προτείνω να αλλάξουμε κάποια στοιχεία της πρότασης. Είχα ήδη την ευκαιρία να μιλήσω για δύο σημεία στον Επίτροπο και φάνηκε ότι δεν είναι όλος όλο εχθρικός πρότασής προτάσεις μου. Ποιε είναι αυτές. Η πρώτη πρότασή μου είναι η εξής. Και μάλιστα στη γνωμοδότηση που διαβάσαμε από την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ, διαβάζουμε ότι θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής του κειμένου να μην έχουμε μια προσέγγιση όπου θα βασιζόμαστε στη θέληση του παραγωγού ή του εκδότη του προϊόντος, αλλά να μπούμε στη θέση του καταναλωτή. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, πρέπει να προκρίνουμε αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στον καταναλωτή που είναι είτε επενδυτής είτε αποταμιευτής να βρίσκεται μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σαφές περιβάλλον, και εκεί να κάνει τις επιλογές του. Εγώ ορμόμαι από την πεποίθηση ότι ο καταναλωτής ε, επιλέγει την επενδυτική του στρατηγική τα για τα θεσμοποιημένα προϊόντα είτε όχι, ανάλογα με τη φύση του δικού τους ας πούμε κινήτρου, είτε έχει, θέλει να κάνει επένδυση είτε αποταμίευση, έπειτα του συνομιλητή του, βασίζεται ε, στην εμπιστοσύνη που έχει στον ε, συνομιλητή του και δεύτερον στη φορολογία του επενδυτικού προϊόντος που θέλει να αγοράσει. Λοιπόν, για αυτά τα τρία θέματα και το πεδίο εφαρμογής. Ε, για την ανάγκη να υπάρχει αυτό το βασικό έγγραφο πληροφοριών, προτείνω να το διευρύνουμε και να μην περιοριστούμε στα δεσμοποιημένα προϊόντα ή στα προϊόντα άγνωστη απόδοσης, αλλά να το διευρύνουμε σε όλα τα επενδυτικά ή αποταμιευτικά προϊόντα χωρίς εξαίρεση. Δηλαδή, από αυτή την πρόταση καλύπτονται και οι μετοχές και τα αποταμιευτικά προϊόντα βάση επιτοκίου συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ομολόγων, οι προθεσμιακοί τραπεζικοί λογαριασμοί και η ασφάλεια ζωή. Όταν παρουσίασα το κείμενο μου στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, Είπα ότι ένας από τους λόγους που προτείνω κάτι τέτοιο είναι ότι φοβάμαι ότι στην νομοθεσία θα προωθήσουμε τα πιο περίπλοκα προϊόντα όπου έχουμε προσπελάσιμη πληροφορία, απλή πληροφορία εις, βάρον, εις βάρος ε, προϊόντων που δεν καλύπτονται από αυτή την νομοθεσία και λένε ότι επειδή είναι πιο απλά αυτά τα προϊόντα δεν προβλέπουμε για αυτά αυτό το βασικό έγγραφο πληροφοριών. Και έτσι δεν ενημερώνουμε τον καταναλωτή. Στο κείμενο τη Κομισιόν υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, όπου λέγεται ότι αυτό το έγγραφο πληροφοριών δεν είναι εμπορικό κείμενο. Ίσως με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε διαφήμιση έτσι των λεγόμενων περίπλοκων προϊόντων. Για να έχουμε συγκρίσιμη διαφήμιση, ξεκάθαρη διαφήμιση, για να έχουμε σωστές πληροφορίες, πρέπει να κάνουμε αυτό που προτείνω εγώ. Για τη φορολογία. Το είπα εισαγωγικά. Για μένα είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Αν είμαστε σοβαροί με τις προτάσεις αυτές και αν δεν θέλουμε απλώς να κάνουμε διαφήμιση των πιο περίπλοκων χρηματιστηριακών προϊόντων, ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει τη φορολογία που θα του επιβληθεί. Νομίζω ότι και οι παραγωγοί μπορούν σε αυτό το έγγραφο πληροφοριών να βάλουν, αν θέλουν, για τη φορολογία αυτών των προϊόντων στις διάφορες χώρες όπου διανέμουν το προϊόν. Για λόγους απλούστευσης, κανένα πρόβλημα αυτό να το αποφασίζει ο παραγωγός. Αλλιώς, όμως, θα πρέπει ο διανομέας να αποφασίσει ε, πώς θα εγγράψει με συνοπτικό τρόπο πληροφορίες για τη φορολογία των προϊόντων αυτών. Φυσικά δεν θέλουμε να υπολογίσουμε τι φόρο θα πληρώσετε. Αλλά να δείτε, ε, να σας πούμε απλά πράγματα. Η ε, υπόκειστε στο ΦΠΑ, στην ε, παρακράτηση στην πηγή, σε τι είδου φορολογία, εν όλα αυτά για ενημέρωση του καταναλωτή. Επίσης, οι δείκτες κινδύνου, σημαντικό στοιχείο. τα ενδεικτικά σενάρια μελλοντικών επιδόσεων βάσει ανάλυσης πολλαπλών συντελεστών π.χ. κίνδυνη αντισυμβαλόμενου προτιμώνται έναντι του δείκτη κινδύνου που βασίζεται στο ιστορικό επιδόσεων. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν δεν είναι σίγουρα θα συμβούν και αύριο. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 22, πρόκειται για μία πρόταση, για μία διαδικασία έγκρισης του συνόλου του εγγράφου θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα είδους stress test ε, που θα το διαχειρίζεται ο παραγωγός. Νομίζω ότι αυτό το σημείο θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Τέταρτος άξονες είναι ε, οι ευθύνε και οι κυρώσεις. Έχω ήδη πει δύο λόγια. Σας προτείνω και ελπίζω να με ακολουθήσει η πλειοψηφία της Επιτροπής, να ενισχύσουμε τις αρχές ε, της των εποπτικών ευρωπαϊκών αρχών. Αυτό είναι και ο στόχος της τροπολογίας 44 που εισαγάγει ένα κεφάλαιο 2α στην πρόταση που επιτρέπει να για τις ΕΙΟΠΑ ε, να δώσουμε τις εξουσίες στην ΕΣΜΑ ούτως ώστε να μπορεί να παρέμβει αυτή η αρχή για τα επενδυτικά προϊόντα λιανεμπορίου και για να περιορίζει, αν χρειαστεί, την διανομή τους ή για να απαγορεύσει τη διανομή τους στο βαθμό που θα παρουσίαζαν ρογμές και κινδύνους. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, πιστεύουμε ότι ο κατάλογος δεν, πρέπει, δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητικός, αλλά όλα όσα έχουν σαν σκοπό να απαγορεύσουν τη διαφήμιση αυτών των κυρώσεων δεν είναι σοβαρά. Η ιδέα της Επιτροπής είναι ότι υπάρχει συστημικός κίνδυνος όταν λέμε ότι το προϊόν είναι τοξικό. Αν αυτά τα προϊόντα λιανεμπορίου θέλουν να διανεμηθούν σε ένα ευρύ κοινό και αν παρουσιάζουν ένα κίνδυνο τοξικότητας τέτοιο που να θέτει να αμφιβόλο την ισορροπία των χρηματαγορών, των ε, χρηματοπιστών αγορών, τότε καλό θα ήταν να το γνωρίζει το ευρύ κοινό το συντομότερο δυνατόν. Γιατί αλλιώς πώς μπορούμε να αποτρέψουμε κάποιους από αθέμητες ε, πρακτικές και από απάτες. Πέμπτος και πρώτο τελευταίο άξονα του κειμένου είναι όλος αφορούν τους, α, τις πληροφορίες για τους επενδυτές σε ό,τι αφορά τον προορισμό αυτών των χρημάτων. Δηλαδή, οι περισσότεροι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν πού πάνε αυτά τα λεφτά, α, τα χρησιμοποιεί ο παραγωγός για να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία και ποιους τομείς της ή για να κάνει απλή κερδοσκοπία ο υπεύθυνο καταναλωτή θα πρέπει να ενεργεί έτσι. Και αυτό θα πρέπει να το υποβοηθήσουμε μέσω διαφανών πληροφοριακών στοιχείων. Επίση, η σχέση αυτού του κειμένου με άλλα κείμενα, με άλλου κανονισμού που συνδέονται. Εδώ ευχαριστώ τη γραμματεία της Επιτροπής μας που μου επέτρεψε να κάνω μια γραφική παράσταση που προσαρτάται στο σχέδιο αυτό της ε, έκθεσης που λέει ποια είναι η δομή μέσα στην οποία εντάσσεται αυτό το κείμενο, καλό να την έχουμε υπόψη μας, στο μηχανισμό της Κομισιόν προβλέπεται μία σύνδεση με την αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ. Ξέρετε ότι για τα ΟΣΕΚΑ η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιβάλλει ένα έγγραφο αντίστοιχο με το βασικό αυτό δικό μας πληροφοριακό έγγραφο. Αλλά, αλλά το όνομα διαφέρει κατά τη και προτείνει να έχουμε ένα περιθώριο πέντε χρόνων για να υλοποιήσουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Εγώ θεωρώ ότι πέντε χρόνια είναι μεγάλο φωνικό διάστημα και θα πρέπει να μειωθεί σε τρία χρόνια. Επίσης, αν διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και στις μετοχές, θα πρέπει να οργανώσουμε το πέρασμα ε, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση της οδηγίας προσπέκτους. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα για τους εμπειρογνώμονες και τους αναλυτές, αναλυτές ε, Standard Poor's για τους, και τους φίλους τους εκεί. Ε, Μιλάμε για ένα μικρό φυλάδιο 15 σελίδων που από ό,τι μου λένε είναι σχεδόν άχρηστο. Ίσως θα πρέπει να πάμε πιο πέρα από αυτά που προτείνω στο κείμενο για να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε το πέρασμα από τη μια υποχρέωση στην άλλη. Θα πρέπει, πάση περιπτώσει, να συνδυάσουμε τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε το κείμενο που εκπονεί ο Βέρνερ για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Επίσης, αναφέρθηκα ήδη στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, η οποία δεν αναφέρεται στο κεφάλαιο 3 για τις προσφυγές, συνεργασία και διεκδικήσεις, ενώ σε αυτό το σημείο σχετικές προτάσεις της ΣΥΜΚΟ θα μπορούσαν να ενταχθούν και να είναι επωφελή για, ε, για το κείμενό μα. Αλλά νομίζω ότι ο εισηγητής τη έχει σκοπό να ασχοληθεί με αυτά ε, σε επίπεδο τροπολογιών. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε που μου επιτρέψατε να παρουσιάσω την ε, έκθεσή μου. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα έχουμε τι συνδυασμένε δυνάμει του Ευρωπαϊκού Γενομένου που συνομώθησαν αντίον μα το, το Eurostar το, το, το χιόνι, όλα αυτά. Την ώρα που άγορευε η περβόνος και τώρα η εισηγήτρια. Ποιητικά είναι. πάνω δύο θέματα όσον αφορά τη, τη γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων που αναφέραμε προηγουμένω, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ότι δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά αυτού του είδου ε, της, της, ε, για τις επενδύσεις. Επίσης η συγκρισιμότητα είναι το άλλο πρόβλημα μεταξύ διαφορετικών προϊόντων. Για τον καταναλωτή. Επομένως, πρώτα απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε υπάρχει διαφάνεια. Και άλλο ένα θέμα το οποίο θέλω να σχολιάσω δεν αφορά μόνο αυτή τη δέσμη των δεδομένων είναι το ότι ο ίδιος ο κίνδυνος αφορά τη δυνατότητα του επενδυτού να καταλάβει τι κίνδυνο, τι ρίσκο λαμβάνει. Και, την άλλη μεριά, Ακόμα και το να διατηρήσει την αξία, του, την αξία της επένδυση και αυτό συνιστά ένα, έναν κίνδυνο να, επομένω, ποια είναι η πολυπλοκότητα και ποιο είναι ο κίνδυνο για τον επενδυτή να χάσει το κεφαλαίο του. Επίση, και εδώ έχουμε θέμα προστασία του καταναλωτού, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη και αυτό θα πρέπει να είναι η αφετηρία τέτοια νομοθεσία. Τώρα, παιδί εφαρμογή, διεύρυνσή του να καλύψουμε και άλλου είδου επενδύσει. Υπάρχει δεσταγμό όσον αφορά την κάλυψη των καταθέσεων. Ίσως είναι δόκιμη η λύση που είχε υιοθετηθεί για τη μύθιν. Τώρα έχουμε τα προϊόντα. Να δούμε πώς θα τα καλύψουμε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα σύγκριση μου. Και να υπάρχει κάποιο κατοχύρωση, εξασφάλιση του κεφαλαίου. Επίσης, το πούμε αυτό όταν φτάσουμε στο σώμα του νομοθετήματος για τις διαφορετικές μορφές ανάλυση του κόστους. Για το ΣΟΣΕΚΑ. Δεν ξέρω αν ε, αυτό το, το ΒΕΠ αυτό αν είναι καλή ιδέα. Γιατί το θέμα είναι τι τι είδους επενδυτές έχουμε να κάνουμε. Έχουμε επενδυτές retail ή όχι. Είναι περίπλοκα τα προϊόντα. Και οι κίνδυνοι επίσης. Οπότε ένα τέτοιο μικροεπενδυτή, ίσω να μην είναι στέση να καταλάβει του κινδύνους. Και ίσως τον ωφελεί το τι κατοχήρωση υπάρχει μέσω των διαφορετικών ε, δελτίων και γράφων πληροφοριών. Τέλο θα πρέπει και το ΒΕΠ να καλύπτει και τους τέτοιου ε, ε, τέτοιους Τώρα, Θα πρέπει επομένω να μπορεί να υπάρχει χρησιμότητα των κινδύνων. Και να λαμβάνει την υπόψη και η διάσταση της μόχλευσης του κάθε προϊόντος. Συμφωνώ με την εισηγήτρια σε όλο το τόσο δύσκολο θέμα του ποιος, ποιος είναι ο δείκτης αντιστάθμισης του κινδύνου. Γιατί εδώ ελαχεύουν κίνδυνοι για τους ε, επενδυτές. Άρα για το μέλλον ίσως είναι σωστό να έχουμε κάποιο είδους πολυεπίπεδες, πολύπλευρες αναλύσεις. Πώς σχετίζεται αυτό το νομοθέτημα με την άλλη που αφορά το, το δελτίο, το ενημερωτικό. Πρόκειται για κάτι το οποίο σωρευτικά βαρύνει. Άρα θα πρέπει το Κοινοβούλιο εδώ να επιμείνει ότι όλες, ε, όλα αυτά τα σχετικά νομοθετήματα να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. των αρχών ε, και το θέμα της ευθύνης αλλά και των κυρώσεων. Να δούμε επίσης τι γίνεται με τον κανονισμό των αλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών. Όταν επομένω υπάρχει κάποιο είδου εναλλακτική κάποια διαιτησία, κάποιο εναλλακτικό τρόπο επίλυση των διαφορών, θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα νομικά δεσμευτικό. Και σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Είμαι σκιώτη εξ ονόματο τη Άλντε. Οπότε θα μιλήσω για κάποια από τα ζητήματα που αναφέρατε. Σα ευχαριστούμε, Περβάν, για το σχέδιο που μα υπέβαλε. Νομίζω ότι πολλά περιλαμβάνει, πολλά περιλαμβάνει με τα οποία συμφωνώ. και την κυρία Πιτικάνεν που ακούσαμε. Ε, θεωρώ ότι είμαι πολλά σύμφωνα από αυτά που αναφέρατε και πραγματικά ανυπομονώ να σημειώσουμε μία πρόοδο. Εγώ θα ήθελα να πετύχουμε πιο πολλά και όχι πιο λίγα, γιατί θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό σε σχέση με τις αρχικές φιλοδοξίες. Ξέρουμε όλοι ότι το Κοινοβούλιο κανονικά είναι το όργανο όπου διατυπώνονται πιο μεγάλες φιλοδοξίες. Τέσσερα σημεία θα αναφέρω σήμερα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ευθύνη για την παραγωγή του έγγραφου αυτού του βασικού. Δεύτερον, ε, δείκτες ε, κινδύνου και τέλος για το κόστος. Σε ό,τι αφορά την ευθύνη για την σύνταξη αυτού του βασικού εγγράφου, είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί καταρχάς θέλω να είναι απλό το έγγραφο αυτό προκειμένου να ξέρει ο επενδυτής σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθεί και ποιος είναι υπεύθυνο, αλλά εκ παραλλήλου σε ό,τι αφορά τον διανομέα, ίσως αυτός να είναι ο, το, ο πιο χαμηλός συντολεστής. Και τελικά αυτός που να έχει τα πιο πολλά χρήματα και που να αξίζει τον κόπο να τον ε, μηνύσει κανείς, να είναι ο παραγωγός. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να βρούμε κάποια κοινή ευθύνη, όσο είναι σαφές ποιο θα είναι το μείγμα. Να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο γιατί και ποιος τελικά έχει την ευθύνη γιατί, σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά από πλευράς περιεχομένου τώρα σε ό,τι αφορά το βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτά που είπε και η ΣΕΡΠΑ, που ενδεχομένω να περιλαμβάνει και άλλε πληροφορίε κτλ. Ενδεχομένω αυτό να επιτευχθεί αρκεί να μην είναι πάρα πολύ περίπλοκο και να μην έχει εξαιρέσει. Ίσως θα μπορούσαν να υπάρχουν αναφορές σε άλλες νομοθεσίες για να μην ξανά αναγκαστούμε να τις ξανααναφέρουμε. Αλλά ασφαλώς δεν μπορούν να υπάρχουν και διαρκείς αναφορές. Αν δείξουμε την απαραίτητη προσοχή, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες περιορισμένες αναφορές για να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκολίες. Τώρα για τους ε, δείκτες κινδύνου. Συμφωνώ και με τις ε, δύο προλαλήσεις δεν ε, μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στο ιστορικό επιδόσεων. Ξέρουμε τι σφάλματα ενέχονται. Και ακόμα και οι μελλοντικοί δείκτες συχνά βασίζονται στις ε, επιδόσεις του παρελθόντος. Άρα θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρχει και αξιολόγηση κινδύνου αλλά και κάποια αριθμητικά στοιχεία. Δεν νομίζω ότι η αναφορά αυτή του κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνει υπερβολικά σχόλια σε ό,τι αφορά εξαιρέσει και αποποίηση ευθύνη κτλ. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται κάποιο απλό περιεχόμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, καταλαβαίνω και θέλω να επεκταθεί για να υπάρχουν ίσοι όροι για όλου στο βαθμό του δυνατού. και θα πρέπει να προσέχουμε να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε, ώστε τελικά να μην καταστεί αδύνατο το εγχείρημα αυτή. Αλλά όπως σας είπα, συμφωνώ να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή και σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που καλύπτει, αλλά και σε ό,τι αφορά του τι φιλοδοξούμε να καλύψουμε, τι άλλο ε, ενδιαφέρει τον επενδυτή. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί το στόχο μας. Και ένας από τους τομείς που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ είναι τα τέλη και οι αμοιβέ. Σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς για την επιβολή προμηθειών, Έχουμε πρόσφατες ε, εμπειρίες στο Ενωμένο Βασίλειο σε περίπτωση απαγόρευσης ε, επιβολής προμηθειών. Αναφέρθηκαν σχετικά στους Financial Times για το ποιες ε, χρεώσεις εξετάζουν τώρα να επιβάλλουν οι τράπεζες πέρα από την ωραία αυτή χρέωση. ποσοστά, 2,5%. Πράγματα τα οποία είναι τελείως ε, παράλογα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ακολουθούν το Ολλανδικό παράδειγμα, όπου απαγορεύονται οι ποσοστίες προμήθειες. Δεν έχω αντίρρηση να επιβάλλονται κάποιες ε, οριές χρεώσεις λογικές. αλλά να δούμε τι χρεώνουν για παράδειγμα, και η παροχή συμβουλών σε τοπικό επίπεδο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι οι, ε, οι επενδυτικοί σύμβουλοι έχουν κάτι κατ' ουσία διαφορετικό. Να δούμε λοιπόν στο MIFID σε ό,τι αφορά θέματα αποποίησης ευθύνεις, να δούμε κατά πόσον μπορούμε να κοιτάξουμε και θέματα περιορισμών. Μπορεί να μην είναι στο σημείο αυτό, αλλά Πρόκειται για μια νομοθεσία η οποία προχωρά μια εποχή που κάτι άλλο ε, είναι μια εποχή που παρουσιάζεται ένα πρόβλημα και γι' αυτό λοιπόν δεν θα έπρεπε να το αφήσουμε το πρόβλημα αυτό να επιδεινωθεί περαιτέρω. Και να περάσω τώρα στο Φιλίπ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη θέση του Σβέν. Και θα μιλήσω στα γαλλικά. Κυρία Συγήτρια, με μεγάλη χαρά σας αναγγέλω ότι οι πράσινοι εκτιμούν πολύ την έκθεση που καταθέσατε. Ας σοβαρευτούμε τώρα. Το πρώτο σημείο που μας με το οποίο συμφωνούμε. Τι λέτε, γίνεται ένας διάλογος εκτός μικροφώνου που δεν ακούμε. Το πρώτο σημείο λοιπόν που μας αρέσει είναι ότι προσπαθείτε όλα τα προϊόντα να τα βάλετε στην ίδια ε, κατηγορία, α, ούτως ώστε να είναι όλα προσπελάσιμα από τον επενδυτή και τον καταναλωτή. Ας μην μιλάμε για επενδυτές, γιατί επενδυτής είναι μεγάλη λέξη, να πούμε αποταμιευτής. Με αυτό λοιπόν το πρώτο συμφωνούμε. Οι Σάρον και άλλοι είπαν ότι θα πρέπει να βασιστούμε ε, και σε άλλους δείκτες, πέρα από τον δείκτη ιστορικών επιδόσεων. Υπάρχουν δείκτες πιο ακριβείς για να δούμε ποιοι είναι οι διάφοροι κίνδυνοι της αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλόμενου κτλ. Σε ό,τι αφορά τα τέλη και τις προμήθειες που χρεώνουν οι ενδιάμεσοι, από τη μία βεβαίως χρειάζεται διαφάνεια, αλλά και εγώ είμαι ρεαλιστής όπως και Σάρων. Είναι ο άσος μας, ο άσος που κρύβουμε στο μανίκι για να μπορέσουμε να βάλουμε λίγη τάξη σε αυτόν τον κόσμο των τεράτων, των λεόντων. Επίσης όλα αυτά που ζητάς από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για την προστασία των επενδυτών είναι σωστά συχνά η εποπτεία είναι ο φτωχό συγγενή. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση λοιπόν στις ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας, θετικό αυτό, μπορούμε να το στηρίξουμε. Όπως είπες, ε, Περβάνς, οι μικροεπενδυτές και οι αποταμιευτές δεν θέλουν μόνο τη σίγουρη αποταμίευση και επένδυση, αλλά τους ενδιαφέρει να μάθουμε και τι γίνεται, τι κάνουμε εμείς με, το, με τα χρήματά τους. Αυτό που λείπει από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι σίγουρα κριτήρια για την βιώσιμη επένδυση. Ακόμα και οι πιο σίγουρες τράπεζες, ακόμα και η Deutsche Bank, ε, έχουν εκεί πέρα μυστικές μαύρες επενδύσεις. Καλό είναι να υπάρχουν λοιπόν ενιαία κριτήρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι είναι βιώσιμη επένδυση ή μη βιώσιμη φυσικά και το ανάποδο. Επίσης, προτείνουμε τροπολογίες που σκοπό έχουν να αυξήσουν τον ανταγωνισμό και, την, τον ανταγωνισμό των γνωμοδοτήσεων που λαμβάνουν οι επενδυτές και να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να περιορίσουμε στο απόλυτα αναγκαίο τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των παραγωγών αυτών των επενδυτικών προϊόντων και των ενδιαμέσων. Γιατί συχνά ο καταναλωτής την πληρώνει. Αυτά νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Θα, θα αναγκαστώ να φύγω γιατί η σύζυγός με περιμένει μέσα στο κρύο. Σας ευχαριστώ. Από το γύρο Στάρ, ε, ο συνάδελφος που ήταν μαζί μου, ο κύριος Καμάλ. Ναι, ναι, ναι. Και φτάσατε μάλιστα και πρώτοι. Και καταλαβαίνω και τα προβλήματα τα συζυγικά που αντιμετωπίζει ο Φιλίπ. Δεν προσβάλλομαι που φεύγει. Mm όπως όλοι οι συνάδελφοι, υποστηρίζουμε τα θέματα διαφάνειας, θέματα ε, ανάληψης των ευθυνών από τον κλάδο και χαιρόμαστε λοιπόν που υπάρχει μια τέτοια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να πω ότι προσωπικά ε, δεν έχω καταλήξει στο ποιος διαβάζει αυτό το βασικό έγγραφο πληροφοριών, μιλώντας και με μέλη ενώσεων καταναλωτών, κάποιοι μα είπαν ότι ναι, ναι, ναι, το διαβάζω. Άλλοι μα είπαν ότι κοιτάξτε δεν το διαβάζω, κοιτάω μόνο τι μου λέει ο αναλυτή μου. Και να σας πω ότι και εγώ δεν διαβάζω και σχετικά έγγραφα. Ενώ διαβάζω σχετική ανάλυση από άλλους. Αυτό το κάνω εγώ προσωπικά ως επενδυτής. Υπάρχει αυτό το βασικό έγγραφο πληροφοριών. Καλό είναι να βασιστούμε σε αυτό, να υπάρχουν κάποια ελάχιστα πρότυπα, αλλά να βεβαιωθούμε ότι δεν θα γίνει πιο περίπλοκο. Να σας ε, μιλήσω τώρα για τους κανόνες του MIFID. Υποστηρίζουμε όλοι ασφαλώς ε, το έργο του Κοινοβουλίου για τη MIFID σε ό,τι αφορά σχετικά, τις σχετικές διατάξεις. Να δούμε όμως πώς θα εφαρμόσουμε το MIFID. Και ποιος είναι υπεύθυνο για την ε, κατάρτιση των πληροφοριών. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ε, των ε, ευθυνών μεταξύ του, του παραγωγού και του διανομέα. Αν θα μπορούσαμε να το διευκρινίσουμε το θέμα αυτό, ίσως θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε και κάποιες από τις ανησυχίε που εκφράστηκαν από την εισηγήτρια. Επίσης, η εισηγήτρια αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή και σε άλλα επενδυτικά προϊόντα. Με μία εξαίρεση. Σύμφωνο απόλυτα. Θεωρώ ότι ακόμα και βασικά τραπεζικά προϊόντα ε, δεν γίνονται κανονικά από τον καταναλωτή. Βάζουν τα λεφτά τους στην τράπεζα αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, μεταξύ στους τραπεζικούς λογαριασμών. Άρα, να τα εξηγήσουμε όλα αυτά στον καταναλωτή. Αλλά να κατανοήσουμε και γιατί οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασίστηκε στους προκατόχους και στους συμβούλους ε, των αρχών που όρισαν σχετικά όρια. Και εγώ το σκέφτομαι ακόμα για το πόσο θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή. Μήπω θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. και να δούμε τι περιλαμβάνει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση. Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικό ούτε σε θέματα λιανικού γενικής πώλησης τέτοιων επενδυτικών προϊόντων, ούτε σε θέματα τραπεζικών υπηρεσιών. Και ξέρω, κυρία Μπερές, ότι είσαστε πολύ ανοιχτοί στη συζήτηση και συμφωνούμε σε διάφορες ε, ιδέες. Άρα, αν υπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας και με τους άλλους συζήτητες. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Κανείς ε, από την ΚΟΕ. Όχι. Κανείς άλλος θέλει το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν. Άρα, Περβάνς, έχεις το λόγο. Did you want the commission? Μήπως ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περβάν says you can have the floor for Τίλμαν, η Περβάν λέει ότι μπορείς να πάρεις το λόγο για λίγο. Αλλά 6.30 ολοκληρώνουμε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε και εμάς το λόγο. Παρότι για λίγο. εκπροσωπώ την Κομισιόν και είμαστε τεχνοκράτες στην Κομισιόν. Θα κάνω λοιπόν κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις για τα στοιχεία της έκθεσης. Καταρχάς υποστηρίζουμε την ιδέα ότι στα επενδυτικά προϊόντα αυτά είναι ε, προϊόντα που ενισχύουν την πραγματική οικονομία. Τα κερδοσκοπικά προϊόντα δεν σημαίνει ότι δεν είναι επενδυτικά προϊόντα αλλά δεν είναι επενδυτικά προϊόντα που θέλουμε να ενισχύσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα σε ένα επενδυτικό προϊόν και σε ένα κερδοσκοπικό επενδυτικό προϊόν. Αν αγοράσει ένα future ή ένα παράγωγο, προφανώς κάνεις ε, επένδυση. Γιατί όταν ε, αυξάνεται η αξία του, ε, τότε μου πληρώνεται μία υπεραξία. Έχουμε λοιπόν ένα επενδυτικό προϊόν Έχουμε και μια ισχυρή διάσταση κερδοσκοπίας ε, στα future. Ε, και αν θέλουμε να κάνουμε διάκριση στον κανονισμό ανάμεσα σε αυτά, και εδώ να το πω ότι είναι κανονισμός, πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στα επενδυτικά προϊόντα και στα κερδοσκοπικά επενδυτικά προϊόντα και πρέπει να κάνουμε μία δοκιμία ανάμεσα στις δύο κατηγορίες, ένα τεστ. Δεν βρήκαμε την διαχωριστική γραμμή. Χρησιμοποίησαμε έναν ουδέτερο όρο γιατί δεν ξέρουμε πού σταματάει η επένδυση και πού αρχίζει η κερδοσκοπία. Για το πεδίο εφαρμογή καταλαβαίνουμε τη φιλοδοξία που εκφράζουν οι ευρωβουλευτέ, την υποστηρίζουμε. Αυτό που πρέπει να επιλύσουμε είναι ότι δεν έχουμε πια ένα παραγωγό προϊόντων, και δεν έχουμε έναν απλό εκδότη. Δεν έχουμε μια τράπεζα η οποία φτιάχνει ένα προϊόν, ας πούμε. Ε, δεν είναι απλά θέματα μόνο μετοχών ή ομολόγων. Ε, επομένως και μια ε, εταιρεία θα πρέπει να εκδίδει ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών και France Telecom. Ε, ανεξάρτητα από το αν, πρόκειται, αν το προϊόν είναι ομόλογα, μετοχές κτλ. Επίσης, η βελγική κυβέρνηση τον εκδίδει ομόλογα στους ε, μικροεπενδυτές. θα πρέπει επίσης να συντάσει ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών και η κυβέρνηση θα πρέπει να μιλάει για τον κίνδυνο ε, σε επένδυση στο βελγικό χρέος, σε αντιδιαστολή με άλλα χρέη. Και αυτό θα ήταν πολύ ε, λεπτό και επικίνδυνο. Πώ συγκρίνει η βελική κυβέρνηση το χρέο σε σχέση με τα άλλα εθνικά χρέη και αυτό θα πρέπει να απεικονίζεται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών. Η μορφή του ΒΕΠ επίσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτή την ειδική κατάσταση. Ε, μπορούμε να έχουμε διαφορετικά ενημερωτικά στοιχεία ε, σε περίπτωση που εκδίδει ας πούμε, η κυβέρνηση αντιδιαστολή με μία επιχείρηση. Ε, ή σε περίπτωση που έχουμε ας πούμε ένα επενδυτικό ταμείο ή μια τράπεζα. Γιατί αν έχουμε επενδυτικό ταμείο αυτό δίνει τελείως άλλες πληροφορίες από την περίπτωση που έχουμε άμεσο ε, εκδότη. Επομένως θα πρέπει το ΒΕΠ να προσαρμόζεται αναλόγως στο ποιος εκδίδει το προϊόν. Σημείο 3. Ε, διαφοροποίηση ανάμεσα στους παραγωγούς και στους ε, διανομή. Η φιλοσοφία είναι ότι ο παραγωγός είναι ο βασικός υπεύθυνος για την έκδοση του web. Γιατί αυτός ξέρει πώς διαρθώνεται το προϊόν, ξέρει ποιο είναι το προφίλ επιδόσεων και πώς υπολογίζεται, ποια είναι τα στοιχεία που πακετάρει σε αυτό το πακεταρισμένο προϊόν. Ο διανομέας μας στην ο διανομέας ε, στη δική μας φιλοσοφία είναι υπεύθυνο για τη διανομή του ΒΕΠ. Δηλαδή θα ήταν υπεύθυνο σε περίπτωση που δεν έδινε το έγγραφο αυτό πριν από την πώληση του προϊόντος. Αλλά δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο του εγγράφου. Γιατί συχνά δεν έχει καμία σχέση με το έγγραφο, δεν καταλαβαίνει ε, καθόλου αυτό το προϊόν και απλώ το διανέμει αυτό το προϊόν. Δεν το φτιάχνει αυτό το προϊόν. Ε, τώρα έχουμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα ε, διάταξη όπου είναι συνυπεύθυνο ο διανομέας με μια α, κοινή και καθολοκληρίαν ε, εγγύηση. Ε, συγγνώμη, συνευθύνη. Αν έχουμε τώρα άμεση έκδοση εδώ, τότε ο διανομέας ξαφνικά παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο γιατί έχουμε μια πλειάδα εταιριών που θα πρέπει να εκδίδουν το ΒΕΠ, ακόμα και κυβερνητικοί φορείς, α πούμε, τοπικέ αρχέ κτλ. Ε, και όταν έχουμε όλη αυτή την πλειάδα των παραγωγών προϊόντων εντό αγωγικών, τότε ενδεχομένω ο διανομέα παίζει μεγαλύτερο ρόλο, γιατί αυτό είναι ο ενδιάμεσο που εξηγεί του κινδύνου. Γιατί σε καμία περίπτωση ο παραγωγός αυτή την περίπτωση μπορεί να το κάνει, γιατί υπάρχει άμεση έκδοση. Υπ' αυτή την έννοια, ο ρόλος του διανομέα πρέπει να συζητηθεί περισσότερο και θα πρέπει να δούμε πώς κολλάει στο όλο πλαίσιο διανομές. Αρχικά δεν να το βάλουμε αυτό το στοιχείο, αλλά και λόγω των τεχνικών εμποδίων με τη σύνταξη για το πώς θα συνταχθεί το ΒΕΠ, ε, θέλαμε να είμαστε έτσι, να καλύψουμε τα νότα μας. Ε, θέλαμε λοιπόν να υπάρχει ένα ΒΕΠ μόνο για τα δεσμοποιημένα προϊόντα γιατί ξέρουμε ποιο είναι ο πάροχο χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών, α πούμε, ε, αυτού και μετά να επεκταθούμε στου άμεσου ε, εκδότε. Σε αυτή την περίπτωση που θα επεκταθούμε θα πρέπει τότε το ΒΕΠ να αλλάξει άρδιν και να είναι πολύ πιο φιλόδοξο. Και αυτό σημαίνει πολύ περισσότερη δουλειά. Τέλος, το, υπάρχουν τα συνταξιδοτικά προϊόντα τα οποία δεν τα έχουμε βγάλει, δεν τα έχουμε αποκλείσει από το πεδίο εφαρμογή ρητά. Υπάρχει όμως μια διάταξη που λέει ότι το σχετικό web γιατί, για το τι α, θα πάρω όταν συνταξιοδοτηθώ, αυτό προτείνουμε να διαγραφεί. Αν το συνταξιδοτικό προϊόν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογή, μιλάμε τώρα για ιδιωτικό συνταξιδοτικό ταμείο, τότε οι, οι πληροφορίε στο web είναι πληρώνω, υπάρχει μια αύξηση αναλογιστικής αύξησης των πόρων και το θέμα είναι τι παίρνω τελικά όταν πάρω σύνταξη. Αν συμφωνήσουμε ότι τα ιδιωτικά συνταξιδοτικά ε, ταμεία εντάσσονται εδώ και τα, τα σχετικά προϊόντα, τότε το ΒΕΠ καλύπτει και αυτά τα προϊόντα. Εμείς θέλαμε να, να έχουμε μια έτσι βαθμία προσέγγιση όταν υποβάλαμε το κείμενό μας. μπορούμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή και εκεί. Αλλά θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να το ξαναδούμε το κείμενό μας. Αν, αν και όταν αποφασίσουμε να βάλουμε εδώ και την, τους άμεσους εκδότες. Βεβαίω να δουλέψουμε. Το θέμα είναι αν θα πρέπει να, αν το κοινοβούλιο θέλει να κάνουμε να αποκινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος πάντων καταλαβαίνω όπως και να είναι τι θέλει να πει η Κομισιόν. Ξέχασα κάτι. Εξαρτώμεθα από το επίπεδο 2. Ότι εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση. Πρέπει επίσης να σας πω ότι χαίρομαι που συμφωνούμε σε τόσα σημεία. Να σταθώ σε δύο όμως, γιατί ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι. Πρώτα-πρώτα, η κατανομή της ευθύνης μεταξύ παραγωγού, δημιουργού και διανομής. Θα πρέπει να έχουμε διαστάσεις, διατάξεις που να είναι εύληπτες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι βάσιμο επιχείρημα και να ρυθμίσει αυτό και την φορολογία του προϊόντος στο σύνολο των χρόνων που θα κυκλοφορήσει. Η κύρια ευθύνη θα πρέπει να αποδίδεται στον δημιουργό του προϊόντος. Δηλαδή αν κάποιος επισυνάψει ένα δελτιάκι που θα λέει τα, τις φορολογικές υποχρεώσεις, αυτό δεν αλλάζει την ευθύνη του. Κάτι άλλο τώρα για το πεδίο εφαρμογή. Ναι, πολλές φορές τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα Αν θέλουμε επίση ο κόσμο να ξαναρχίσει να αγοράζει μετοχέ, ε, τότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και να δούμε κατά πόσον εάν η διεύρυνση του πεδίου θα είχε αυτά τα αποτελέσματα επίσης τελευταίο σημείο με τις συντάξεις Είμαι λίστα και γι' αυτό. Δεν πρότεινα να έχουμε εκεί διάμεση του πεδίου εφαρμογή όσον αφορά τι συντάξει. Θα ασχοληθεί πάντω με αυτό η Επιτροπή Ιστορική Αγορά. Για να δούμε ποιοι συνάδελφοι θέλουν αυτό να το κάνουν. Να δούμε αν αυτό θα ρεμιστεί τώρα ή αργότερα που θα υπάρξουν διαπραγματεύσει σχέση με την οριστική θέση που θα, θα υιοθετήσει το Κοινοβούλιο. Οπότε, κατόπιν των όσων είπατε, μπορείτε να υποβάλλετε, να υποβάλλετε σχετικές τροπολογίες, δεν έχω καμία αντίρρηση. Τώρα το, το ποιες θα περάσουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά θα σχολιάσουν. Τέλος για σήμερα. Hey, thank you very much. Uh, now have a deadline for a... Σας ευχαριστούμε. Έχουμε δώσει προθεσμία για τις την 6η ε, Δευτέρα. Και θα τα συζητήσουμε στις 25 ε, Δευτέρα. Και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 26 Τρίτου. Και έτσι θα ακολουθεί θεωρητικά στην Ολομέλεια του Μάιου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Πριν κηρύξουμε την λήξη της εμβριάσεως, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει για την τελευταία ημέρα που ο κύριος Γιούνκερ προεδρεύει το Eurogroup. Είχε έρθει εδώ πριν μια εβδομάδα. Θα μας λείψει και αυτός, το χιούμορ του, η ευθύτη του. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε ο διάδοχός του να ανταποκριθεί στην φήμη του κυρίου Γιούνκερ και στην αξία του. Ενιά η ώρα αύριο θα συνεχίσουμε και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες όσον αφορά την οδηγία για το κοινό σύστημα ε, ΦΠΑ. Ευχαριστούμε.